Να συνεχίσουμε τώρα με τη συνεδρίασή μας και να εξετάσουμε τα εγκάρσια ε, ταμεία υγείας έναντι των βασικών συστημάτων υγείας. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση για τα εγκάρσια ταμεία που εμφανίστηκαν πριν 10 χρόνια περίπου. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις για τα ταμεία αυτά. Ορισμένοι θεωρούν ότι συνεισφέρουν στον κατακαιρματισμό της ε, βοήθειας και ότι εκτρέπουν τις πηγές χρηματοδότησης προς τις ε, συγκεκριμένες ε, ασθένειες της βάρους της στήριξης της ε, υγείας, ενώ άλλοι εκτιμούν ε, ότι έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους και έχουν καταγράψει θεματικά αποτελέσματα. Γι' αυτό σήμερα έχουμε καλέσει προσώπους της Κομισιόν ε, του Παγκόσμιου, Ταμείου, συγγνώμη, του Παγκόσμιου Ταμείου Καταπολέμησης του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελληνοσίας και της ΠΟΗ. Υποδεχόμαστε τον κύριο Ριέρα, ο οποίο είναι διευθυντή τη ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξη, τον κύριο Καζαξίν, εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Ταμείου και την κυρία Βέμπερ Μόσντορφ, διευθύντρια του Γραφείου της Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας της Βρυξέλλες. Για να ξεκινήσουμε, θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Καζάτσκιν, ο οποίος θα μας ε, παρουσιάσει ε, το Παγκόσμιο Ταμείο που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια περίπου. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Ζουλή, που βάλατε το θέμα της υγείας σήμερα στην ημερησία διάταξη της Επιτροπής σας και με καλέσατε να σας απευθυνθώ εκ μέρους του Παγκοσμίου Ταμείου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, οικονομική και πολιτική υποστήριξη στο Παγκοσμίο Ταμείο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχήν, η υγεία είναι ο τομέας της ανάπτυξης, όπου έχουμε σημειώσει θεματική πρόοδο τα τελευταία δεκαέτη, αλλά θα έλεγα ακόμη περισσότερο τα τελευταία πέντε έτη. Αυτά τα τελευταία πέντε δεκαέτη βιώσαμε πρωτοφανή ενεργοποίηση ή κινητοποίηση, αν θέλετε, της ε, κοινωνίας στο Βορρά και στο Νότο, πρωτοφανή πολιτική δέσμευση και για την εξέβρεση των οικονομικών πόρων που ενεργοποιούνται για την υγεία. Θυμηθείτε, το 2001 σχεδόν κανείς με AIDS δεν ε, λάμβανε σε αναπτυσσόμενες χώρες αντιοική θεραπεία, ενώ στα τέλη του 2008 έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα που έχουν πρόσβαση σε θεραπεία για το AIDS, αποτελούν Έχουμε δηλαδή περίπου κάλυψη 40% των όσων είναι σε έκτατη ανάγκη, σε πήγουσα ανάγκη. Και είδαμε τώρα τον αντίκτυπο αυτή τη χρηματοδότηση σε επίπεδο πληθυσμού. Μειώθηκε η θνησιμότητα από AIDS σημαντικά σε πολλέ ε, χώρε με υψηλό άχθο στην Αιθιοπία. Μειώθηκε κατά 60% τα τελευταία πέντε χρόνια και ο αριθμός των νέων ε, HIV μολύσεων μειώνεται σε αρκετές χώρες της υποσαχαρίας Αφρικής. Το 2001 η ελληνοσία ήταν μια παραμελημένη νόσος, ενώ σήμερα τουλάχιστον 10 από τις ε, ε, πλέον και ε, χώρε στην υποσαχαρή Αφρική έχουν αναφέρει μείωση σε νέα κρούσματα ελαιονοσίας ε, και έχουμε μείωση της νησιμότητας των παιδιών από 40, 40 και 80% και η συνολική επικράτηση της εφηματίωσης μειώνεται παγκοσμίω. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι αν διατηρηθούν οι προσπάθειες αυτές και επεκταθούν, τότε υπάρχει πραγματική ευκαιρία να έρθουμε κοντά ή να φτάσουμε τους ε, διάφορους ε, στόχους της χιλιετίας που σχετίζονται με την υγεία. Έχουμε ε, τον στόχο 6 για τα διεθνή πρότυπα και θα έπρεπε να σημειώσουμε και σημαντική πρόοδο για τον στόχο 5 και για τον στόχο 4 για τη θρησιμότητα των μητέρων αν ε, συνεχιστούν οι προσπάθειες στο σημερινό επίπεδο. Η ελληνοσία θα μπορούσε να εξελιχθεί ως πρόβλημα της δημόσιας υγείας στις ε, περισσότερες χώρες όπου εκδηλώνεται και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε το 2015 ένα κόσμο χωρίς θανάτους από ελληνοσία έχουμε ε, τη δυνατότητα μέσω της ε, πρόληψης ε, να προστατεύσουμε πολλούς ανθρώπους από τη μόλυνση του ιού του AIDS και μπορεί να συγκρατήσουμε και την εξάπλωση της φυματίωσης μπορούμε να εξαλείψουμε επίσης την μετάδοση από μητέρα σε παιδί του HIV. Τρίτο πρόεδρε. Το Παγκόσμιο Ταμείο έχει διδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην πρόοδο που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και ο ρόλος του Παγκόσμιου Ταμείου αφορούσε όχι μόνο την άμεση χρηματοδότηση, την εγκάρσια χρηματοδότηση και την, ε, την... χρηματοδότηση ε, στρατηγικών για την πρόληψη, αλλά ταυτόχρονα ενδυνάμωσε τα συστήματα υγείας προκειμένου οι χώρες να μπορέσουν ε, να παραδώσουν, ε, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων. Θα σταθώ σε αυτό το θέμα για το Παγκόσμιο Ταμείο. Το Παγκόσμιο Ταμείο, όπως, μπορούν, ε, όπως μπορεί να θυμάστε, δημιουργήθηκε όταν ε, συνειδητοποιήθηκε στις αρχές ε, του 2000 ε, ότι δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στην επιδημία του AIDS όπως και στη φυματίωση και στην ελωσία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί είχαμε λοιπόν μία πρωτοφανή κρίση ανθρωπιστική και ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ στις Βρυξέλλες μέσω της Μετανατικής Ομάδας Εργασίας το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεπλά σαν ενεργά μετά την έκκληση του Κόφι Ανάν ε, όπως ε, αποκάλεσε την περίπτωση αυτή, είχαμε έναν πόλεμο κατά του AIDS. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποιες από τις κύριες αρχές ε, για το πώς εργαζόμαστε στο Παγκόσμιο Ταμείο. Καταρχήν, το Παγκόσμιο Ταμείο βασίζεται στην συμμετοχή Πρόκειται για έναν οργανισμό λήψη αποφάσεων όπου συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε κάθε επίπεδο από ε, το επίπεδο των χωρών ε, όπου έχουμε τους μηχανισμούς λήψη αποφάσεων από τις οργανώσεις που στέλνουν τα αιτήματα στο Ταμείο μέχρι το Συμβούλιο που έχουμε ισότιμη εκπροσώπηση των δωρητών και των όσων εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές στον τομέα της ανάπτυξης και ε, η συμμετοχή ε, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινοτήτων, του ιδιωτικού τομέα και διάφορων εταίρων είναι πολύ μεγάλη. Όλοι αυτοί από κοινού λαμβάνουν τι αποφάσει. Στο δικό μα συμβούλιο, ο εκπρόσωπο από τι πληγήσει κοινότητε έχει το ίδιο δικαίωμα ψήφου όπω ο εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνεισφέρουν ε, ένα δισεκατομμύριο συνεισφέραν φέτο η ύπα στο Ταμείο. Το δεύτερο είναι το λεγόμενο country ownership, δηλαδή στήριξη ε, των ε, προγραμμάτων του Ταμείου όπου έχουμε τις εθνικές προτεραιότητες. Οι ίδιες οι χώρες ε, βάσει των προτεραιοτήτων τους παίρνουν τις αποφάσεις, μεταφράζουν τις αποφάσεις αυτές σε αιτήματα που τα υποβαλούν στο Ταμείο και γίνεται στη συνέχεια αξιολόγηση της ποιότητάς τους, της επιστημονικής ε, ποιότητας και άλλων πτυχών οι ε, επιστημονική ποιότητα και άλλε εξετάζονται πριν να γίνουν αποδεκτά από το Ταμείο. Επίση, ε, αναλύουμε μόνο ε, προτάσει οι οποίε βασίζονται σε συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Και επίση, έχουμε και ένα μοντέλο για την κατανομή των κονδυλίων που να είναι απόλυτα διαφανές για τους δωρητέ και για του δικαιούχου. Αν πάτε στην ιστοσελίδα μας κάθε εβδομάδα θα δείτε πώς εκταμιεύονται τα κονδύλια και πώς δαπανώνται. Επίσης ε, θα δείτε τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων και των ερευνών που υλοποιεί το Ταμείο. Όπω ε, σας είπα, ήταν τεράστια η πρόοδο που σημειώθηκε. Το Παγκόσμιο Ταμείο έχει ε, τώρα αύξηση πάνω από 90 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το μεγαλύτερο ε, συνεισφέροντα στους στόχους της χιλιετίας ε, για την ανάπτυξη και έχουμε σώσει μέχρι και 5.000 ε, 5 εκατομμύρια ζωές. 3.000 ζωές σώζουμε την ημέρα στον απτυσσόμενο κόσμο. Σε σχέση με την άμεση χρηματοδότηση, οι παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας γίνονται για ε, τρεις, ε, για αυτές τις τρεις νόσους ε, και το Ταμείο είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στα στήματα υγείας. Το 35% των επενδύσεών μας, 35% δηλαδή των 19 δισεκατομμυρίων που έχουν μέχρι τώρα δεσμευτεί, έχουν επενδυθεί στην ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας και στη βελτίωση της διοίκησης, της προμήθειας, της ικανότητας παρακολούθησης, την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην ενδυνάμωση των κοινωνία των πολιτών και των κοινοτήτων. Στην Αιθιοπία, λόγου χάρη, όπου έχουμε το μεγαλύτερο δικαιούχο των πόρων αυτών στην Αφρική, η Αιθιοπία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για το AIDS και την ελληνοσία που λαμβάνει από το Παγκοσμίο Ταμείο για να οικοδομήσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υγείας ε, που ε, έχουμε ε, πρόσθετους εργαζομένους και εκεί συνδυάζεται η υπηρεσία πρόληψης και παροχής ε, φαρμάκων. Έχουμε επίσης βασική υγιεινή πρόληψη και αντισύλληψη. Αυτό στο πλαίσιο των στρατηγικών της μείωσης της φτώχειας. Τέλος, τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από τα ταμεία ε, είναι ε, αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να τα συνδέσουμε με την ε, συγκεκριμένη προσπάθεια που καταβαλούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την περίοδο 2002-2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνιστούν πάνω από το 50% των συνολικών δεσμεύσεων και σφορών στο Παγκόσμιο Ταμείο και αν λάβουμε και τις ορευτικές ε, δεσμεύσεις και σφορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σήμερα ο τέταρτος μεγαλύτερος δωρητής στο Παγκόσμιο Ταμείο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιαπωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τμήμα της παγκοσμίας διακυβέρνησης στο Συμβούλιο μας, αλλά και σε επίπεδο χώρας ε, μέσω των μηχανισμών ε, συντονισμού ε, αναχώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην χάραξη της πολιτικής για την ανάπτυξη. Υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος παγκοσμίω στους σχετικούς με την υγεία στόχους της χιλετίας. Έτσι λοιπόν, εσείς ως βουλευτές και πολίτες θα πρέπει να αισθάνεστε ότι και η επιτυχία του Ταμείου και το μέλλον του Ταμείου είναι και κάτι δικό σας. Έτσι έρχομαι στο τελευταίο τελευταίο σημείο που έχει να κάνει με το 2010. Το 2010 είναι θεμελιώδε έτο για την ανάπτυξη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο κόσμο θα φτάσει στο να το πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τη χιλιετία. Και ρόλο σα εδώ ω ευρωβουλευτέ είναι σε αυτή η διαδικασία. Το 2010 είναι το έτο όπου ο κόσμο θα αναθεωρήσει την πρόοδό του για του στόχου τη χιλιετία. Επίσης είναι το έτος όπου το Παγκόσμιο Ταμείο θα ε, ε όπως ε, κάθε τρία χρόνια θα ζητήσει νέα κονδύλια για, ε, θα λάβει μια χρηματοδότηση για τα έτη 11, 12 και 13. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ανασύσταση των κονδυλίων θα καθορίσει πού θα βρίσκεται ο κόσμος το 2015 σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας σχετικούς με την υγεία. Και ως ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θεμελιώδης ο ρόλος στη διαδικασία αυτή της ε, ανασύστασης ε, του Ταμείου. Η υγεία έχει να κάνει με την ανάπτυξη, η ανάπτυξη έχει να κάνει με τις διεθνεί σχέσεις, με το τι είδους παγκοσμιοποιημένο κόσμο θέλουμε να οικοδομήσουμε και η υγεία λοιπόν είναι ένα ζωτικό πολιτικό ζήτημα. Αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την συνεισφορά τη στο Παγκόσμιο Ταμείο και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το δικό σα ηγετικό ρόλο στα θέματα τη παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη και για την υποστήριξη που έχετε επιδείξει στο Παγκόσμιο Ταμείο και μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στα κράτη-μέλη σα. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Βέμπερ Μόστοροφ για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πρόσκληση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να κάνουμε έναν απολογισμό και να μάθουμε τι ακριβώς έχει λειτουργήσει καλά και τι όχι, τι μένει ακόμη να γίνει κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά και μετά. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με τον ε, προλαλήσαντα συνάδελφο ότι έχει σημειωθεί πολύ πρόοδος και ότι από, από τότε που από το 2005 έχει τετραπλασιαστεί η, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και νομίζουμε ότι αυτό συνιστά μία πρόοδο. Και η υγεία είναι πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πολλές φορές το παρελθόν είχε υποτιμηθεί ως ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά είχε υποτιμηθεί και ως προς τη σημασία της για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οπότε το θέμα δεν είναι τόσο τα εγκάρσια μία σε σχέση με την ε, κύρια φροντίδα. Το θέμα είναι πώς ε, μπορούμε να τα συντονίσουμε με συγκεκριμένα προγράμματα και με πρόοδο στη δημόσια υγεία, ενσωματώνοντας, εθνικέ ε, εθνικές ε, στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και που αντιμετωπίζουν ε, τις κύριες αιτίε της ασφάλεια, της, των ασθενειών, όπως για παράδειγμα ο υποσυτισμός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF ε, έχουν ε, ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για το καθαρισμό του νερού και για τις ε, αποχετεύσεις που νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό τμήμα της δουλειάς μας και μια σημαντική αιτία πολλών ασθενειών. Οπότε θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στους στόχους της χιλιετίας και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Ο 4 και ο 5 με τον 1 για παράδειγμα ή με τον 7. Δηλαδή περιβαλλοντική στόχη της χιλιετίας, ε, νερό και αποχέτευση, όπως επίσης ε, και ο στόχος 8, μετάδοση της τεχνολογίας ε, και φθηνή πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και στα φάρμακα. Πρέπει να δούμε δηλαδή την ευρύτερη εικόνα αν θέλουμε να εξετάσουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει. Και αυτό που θα ήθελα πολύ σύντομα να κάνω είναι να εξηγήσω μερικά σφάλματα που έγιναν και όχι να κατηγορήσω κανέναν για τα σφάλματα αυτά, απλώ να πω ότι υπάρχουν κάποια συστηματικά προβλήματα, κάποιες συστηματικές αδυναμίες. Και θα ήθελα επίσης να δούμε και τις μελλοντικές προκλήσεις. Να δούμε επίσης πώς μπορούμε να επισπεύσουμε την ε, βελτίωση. Αν δούμε για παράδειγμα τον τέταρτο στόχο, ένα, ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι για παράδειγμα η διάρκεια. 1,5 εκατομμύρια στην υποσαχάρια Αφρική και στην, νοτιοανατολική Ασία. Είναι θλιβερό. Γιατί υπάρχουν θεραπείες, υπάρχουν μέσα, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με αποτελεσματικό και όχι πολύ δαπανηρό ε, τρόπο. 1,5 εκατομμύρια, πολύ μεγάλος αριθμός ε, και επίσης έχουμε και 2 εκατομμύρια λόγω της πνευμονίας, θανάτων από πνευμονία είναι κάτι το οποίο δεν έχει επαρκώς εξεταστεί. Ο στόχο 5 γνωρίζετε τα αριθμητικά στοιχεία, δεν υπάρχει λόγο να τα επαναλαμβάνω, αλλά για παράδειγμα για μα αυτό αποτελεί έναν δείκτη υγεία που δείχνει τα μεγαλύτερα χάσματα μεταξύ, τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ε, φτωχών και των πλουσίων και ακόμη βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου λιγότερο από 50% εγγύων γυναικών ε, είχαν τη δυνατότητα τεσσάρων ε, ελέγχων προγεννητικών, 61% μόνο των γυναικών Λοιπόν, ε, υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού και πολύ λίγες ε, ε, επισκέψεις μετά τη γέννηση, κάτι το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με πολλούς άλλους στόχους, όπως για παράδειγμα της ιατρικής περίθαλψης γενικά. Το θέμα τώρα της, την εφηβική εγκυμοσύνη, τα υψηλά επίπεδα, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα σε μερικές χώρες. Έχει αυξηθεί επίσης ε, το ποσοστό της αντισύλληψης σχεδόν σε όλες τις χώρες, αλλά στην ε, δική μας την περιοχή 108 ε, εγκυμοσύνες στις χίλιες και μιλάω για την εφηβική εγκυμοσύνη για τον, την περιοχή που μας απασχολεί εμάς. Είναι ένα υψηλό ποσοστό. Δεν είναι επαρκής ακόμα οι υπηρεσίες ε, ιατρικές ε, για τις ε, έφηβες αυτές, ούτε για τους εφήβους. Αν δούμε ότι 21% για παράδειγμα των εγγύων εξετάζονται για AIDS και 30% των ανδρών, 19% των νέων γυναικών εγνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει ο ιός του AIDS. Αυτό μας δείχνει σαφέστατα ότι χρειαζόμαστε αυτές τις υπηρεσίες ε, οικογενειακού προγραμματισμού και αυτήν την ε, πρόσβαση ε, σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Κάτι ακόμη, κάθε χρόνο 400 εκατομμύρια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ε, καταγράφονται 40% των προγεννητικών ε, θανάτων ε, ακριβώς προκύπτουν από τη μη θεραπεία της σύφυλης. Βλέπετε λοιπόν τι τεράστια που είναι τα ποσοστά. Ας δούμε λοιπόν τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και που τις διαπιστώσαμε μετά από πολλά χρόνια πρόοδου. Βασικές λοιπόν προκλήσεις ε, είναι η ισότητα και τα προβλήματα της ιατρικής, ε, των ιατρικών συστημάτων, ειδικότερα στις ε, φτωχές χώρες. 63% των θεραπείων για την διάρρεια, 54% για σοβαρές λοιμώξεις και 50% για υποστήριξη στο τοκετό. Αν δούμε λοιπόν την πρόοδο στους αναπτυξιακούς ε, στόχους της ε, χιλιετίας, ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων, των ανδρών και των γυναικών και ακόμη και στο πλαίσιο μιας χώρας μεταξύ διαφόρων εθνικών ομάδων υπάρχουν σημαντικές διαφορές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να επισπεύσουμε την πρόοδό μας. Κάτι το οποίο θεωρούμε σημαντικό είναι μεγαλύτερη επένδυση σε αλληλεγγύη και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να προστατευθούν οι δαπάνες για την υγεία των κυβερνήσεων όπως επίσης και των δωρητών. Επίσης, θα θέλαμε να δοθεί περισσότερη προσοχή και να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας ε, με πιο περιεκτικό τρόπο. Δηλαδή όχι μόνο εγκαρσίως, ε, αλλά και ιατρικά προϊόντα, τεχνολογία, εξοπλισμός, ε, ιατρικό προσωπικό, κοινωνική ασφάλιση, συστήματα ενημέρωσης για τα θέματα της υγείας και επίσης να ε, καθίστανται οι χώρες υπεύθυνε για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών. Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η πρόσβαση και ειδικότερα στις ευάλωτες περιοχές και τις ευάλωτες ομάδες με ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχούς, ε, με τους φτωχότερους πληθυσμούς ε, και στις γυναίκες. Εφαρμογή κοινωνικών μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε οικουμενικές υπηρεσίες και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να περάσω στις δυνατότητες που έχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα ε, ζητήματα που συζητούμε ιδιαίτερως εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι η ενίσχυση της διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο χωρών. Αν δούμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και νομίζουμε ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό βήμα, ότι εντός του ε, ΠΟΗ μεταξύ των 193 χωρών υπήρχε σαφή συμφωνία και δέσμευση για ε, τις αρχές αυτές ε, της πρόσβασης ε, σε πρωτογενείς ιατρικές υπηρεσίες, ότι αυτό είναι μια βασική αρχή. Πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για το τι γίνεται στην κάθε χώρα Κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι και οι χώρες ε, αποδέκτες πρέπει να επιτύχουν ε, το 50% ε, του εθνικού εισοδήματος που θα παρέχεται στην προσπάθεια αυτή. Επίσης, πρόσληψη του σωστού προσωπικού. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές προσλαμβάνουμε προσωπικό από την Αφρική, για παράδειγμα. Πρέπει να δούμε επίσης και τους κοινωνικούς παράγοντες. Υπάρχουν ε, συστάσεις ε, στο πλαίσιο των ε, κυβερνητικών φορέων του ΠΟΗ και πρέπει να δούμε τις παγκόσμιες πολιτικές, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλέον ένας παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο για το θέμα αυτό. Μπορούμε να ανταποκριθούμε πλέον σε τέτοιου είδους προκλήσεις ε, μέσω κοινωνικών πολιτικών για παράδειγμα. Ένα λοιπόν πολύ σημαντικό βήμα θα ή, για την βελτίωση της διακυβέρνησης θα ήταν να ενισχύσουμε ε, στρατηγικές και υποδομές ε, των κρατών Στι οποίε απευθυνόμαστε, να τα αναλάβουν οι ίδιε οι χώρες δηλαδή. Αν δούμε για παράδειγμα το μεγαλύτερα, μεγαλύτερα προβλήματα είναι ε, μεταδοτικέ ασθένειε, αλλά υπάρχουν και μη μεταδοτικέ ασθένειε. 33 εκατομμύρια των ε, θάνατοι στι αναπτυσσόμενε χώρε είναι από μη μεταδοτικέ ασθένειε. Επομένω, οι αναπτυσσόμενε χώρε ε, έχουν δύο είδη προβλημάτων. Επιδημιολογικές καταστάσεις, πράγματα τα οποία εμείς ε, στην Ευρώπη τα έχουμε αντιμετωπίσει σε πιο μεγάλες περιόδους μετα, μετάβασης και όμως είναι σημαντικές προκλήσεις σε άλλες χώρες. Επίσης πρέπει να καλύτερη παροχή ε, της ιατρικής φροντίδας ε, και γενικότερα όλες οι προσπάθειες στον ιατρικό τομέα σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι αντικείμενο συντονισμού μεταξύ των χωρών που είναι δωρητές, για παράδειγμα μέσω παγκόσμιων ε, παγκόσμια συνεργασίας και μέσω της πλατφόρμας που ανέφερε ο συνάδελφος προηγουμένως. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ε, πραγματικά δείχνουν αυξανόμενη συγγνώμη, αναγνώριση της ε, κατάστασης του τομέα της υγείας και, ότι, και πόσο σημαντικό είναι να κατέχουν τις υποδομές οι ίδιες οι χώρες ώστε να μπορούν, να, να μπορούν και εκείνες να συμμετέχουν αλλά μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες ε, οπόη έχει γραφεία σε 150 χώρες. Ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται, είμαστε παρόντες στις χώρες αυτές και τις υποστηρίζουμε. Σε σχέση με τις προτάσεις, για παράδειγμα, για το Παγκόσμιο Ταμείο. Έχουμε επίσης τις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές και νομίζω ότι θα έπρεπε πραγματικά να αξιοποιήσουμε πολύ την ευκαιρία αυτή ώστε να είναι πολύ πιο ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ναι. ως ε, θεματοφύλακας αλλά και ως ε, παράγον που προάγει τον τομέα της υγείας. Ε, νομίζουμε λοιπόν ότι αυτά, ήταν τα βήματα που αυτά είναι τα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί και θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ριέρα από τη ΓΑΜΑ Δελτανάπτυξη για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Καταρχήν, ευχαριστώ που καλείτε την Κομισιόν να μοιραστεί μαζί σας τις απόψεις της και να συμμετάσχει στην σημερινή συνεδρίαση. Μετά από την εκπρόσωπο του ΦΑΟ, διορθώνει ο όχι της ΦΑΟ, της ΠΟΗ. Ε, ένα, πολλά θέματα ακούστηκαν ήδη, αλλά να τονίσω κι εγώ κάποια από τα βασικά σημεία που πιστεύω ότι μπορεί να είναι χρήσιμα στη σημερινή συνεδρίαση. Καταρχήν, η Κομισιόν ευχαριστεί για την υποστήριξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ε, ιδρυτικό μέλος της ε, παγκόσμιας ε, χρηματοδότησης συμμετείχε ενεργά από την αρχή και δεν είναι θέμα αριθμητικών στοιχείων αυτό που δείχνει τη συμμετοχή μας, αλλά είπαμε ότι από το 2002 η Κομισιόν μέσω της υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει για πάνω από 800 σχεδόν 900 εκατομμύρια ευρώ που μπήκανε στο Παγκόσμιο Ταμείο. Και όπως ε, υπόθηκε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη ε, αντιπροσωπεύει πάνω από 50% των συμβολών, των συνσφορών στο Παγκόσμιο Ταμείο. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω από την πλευρά της Κομισιόν ότι εμείς όλο και περισσότερο δρούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παγκόσμιο Ταμείο. Συμμετέχουμε στις δραστηριότητε του και στις συμπράξεις του από την πλευρά της Κομισιόν, ειδικά τώρα που έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που μας δεσμεύει να ενισχύσουμε τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό να γίνει με ένα αρμονισμένο τρόπο. Και ειδικά τώρα που γίνονται αλλαγές κλειδιά για το Παγκόσμιο Ταμείο, το έχουμε αναφέρει, το είπε και ο Μισελ την, ε, για το εγχείρημα εμπλουτισμού, ενίσχυσης που είναι αρκετά σημαντικό, αλλά και πέρα από αυτό νομίζω ότι το Παγκόσμιο Ταμείο έχει φτάσει ένα σημείο που θα έπρεπε και με, είτε με το, με το ε, αυτό είτε χωρίς ε, να, είναι, να γίνει πραγματικά μια πολύ συγκεκριμένη και σοβαρή ενδοσκόπηση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι αυτό το έχουμε κάνει στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκπαιδευτικής Γραμματείας, η οποία πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ. γιατί μας επέτρεψε να κάνουμε έναν, μια σαφή ε, σοβαρή ενδοσκόπηση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Επί τη βάση βέβαια των ε, επιτυχιών που έχουν ήδη υπάρξει και που αναφέρθηκαν ήδη πριν από λίγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πλαισιώσουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν στο Παγκόσμιο Ταμείο ε, και μέσω του τέταρτου προγράμματος που θα παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Στο πακέτο λοιπόν αυτό για την ενδιάμεση αναθεώρηση των στόχων της, της χιλιετίας στην Νέα Υόρκη για την παγκόσμια υγεία. Ήδη θα ξέρετε ότι εκτός από το ότι βάζουμε την, θέτουμε, δίνουμε σημασία στα ποσοτικά θέματα, η Κομισιόν θέλει να μελετήσει και το τι θα γίνει στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης επί τη βάση μιας καλύτερης ε, ε, προ... πολιτικής για τους διάφορους τομείς που μας απασχολούν και να έχουμε μια προσέγγιση η οποία θα μπορέσει να έχει μια προσθέμενη αξία. Ελπίζω σύντομα να λάβετε δύο ανακοινώσεις, μία για την παγκόσμια υγεία και μία για την, ασφάλεια, την διατροφική ασφάλεια. Και επίσης θα λάβετε δύο έγγραφα ένα, για, ένα θέμα, για ένα πρόγραμμα δράσης ε, για, για τα δύο φύλλα και ένα έγγραφο για την καλύτερη και περισσότερη εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, και το είπε η Διανέτ, το θέμα της, του εσωτερικού, της εσωτερικής χρηματοδότησης των χωρών που είναι αποδέκτες για, το, για, τους, για την επίτευξη του, των στόχων της χιλιετίας είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει μέσω αυτού του προγράμματος με αυτόν τον τρόπο να, γίνει η, να συνεχιστεί η υποστήριξή μας προς το Παγκόσμιο Ταμείο. Γιατί έτσι μπορούμε να δείξουμε ότι σε ό,τι αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και πέρα από την άμεση ενίσχυση που δίδει η Κομισιόν με τη δική σας συμβολή προς κάποιες χώρες μέσω άμεσων δράσεων και προγραμμάτων. Οι δύο βασικοί παράγοντες των παρεμβάσεων μας στην υγεία είναι η παγκόσμια υγεία και το Παγκόσμιο Ταμείο και δεύτερον οι δράσεις μας μέσω της υποστήριξης ε, του προπολογισμού το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, θεωρούμε ότι σε έναν τομέα όπως είναι η υγεία, αλλά και η εκπαίδευση, όπου τα λειτουργικά κόστη είναι τόσο πολλά, να δώσουμε στις χώρες αυτές ένα πλαίσιο προβλεψιμότητας για τις δυνατότητες που έχουν να συμβάλλουν, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους στους τομείς αυτούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, εμείς πιέζουμε να υπάρξει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον τομέα της υγείας και στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας. Και αυτό έχει να κάνει και με την καλύτερη προβλεψιμότητα και για το δικό μας προπολογισμό, όχι ως αντιστάθμισμα, αλλά ως τμήμα μιας σύμβασης όπου οι χώρες, οι επιλέξιμες θα ανταποκρίνονται στους κοινωνικούς στόχους της ε, χιλιετίας και στις κοινωνικές πολιτικές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και στα πλαίσια των σχέσεων μας με το Παγκόσμιο Ταμείο είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι δύο άξονες της πολιτικής μας ε, θα συγχωνευτούν, θα συνδυαστούν. Πραγματικά έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη μας την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, γιατί δεν υπήρχαν μέχρι τώρα αρκετές συνέργειες και σχέσεις μεταξύ της δικής μας υποστήριξης στον τομέα της ε, υγείας για κάποιες χώρες και της υποστήριξης που ε, στοχοθετούμε μέσω του Παγκοσμίου Ταμείου. Ε, ω προς, το προς την επίτευξη του στόχου λοιπόν αυτού, πέρα από τη συμμετοχή στο Συμβούλιο, ε, έχουμε οργανώσει με έναν αριθμό σεμιναρίων με τις ε, υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες του ε, Παγκοσμίου Ταμείου, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει καλύτερη κατανόηση για τους τρόπους με τους οποίους συλλειτουργούμε. Έχουμε εκδώσει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις αντιπροσωπείες μας για τον τρόπο που μπορούμε να ενισχύσουμε, να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνέργειες και έχουμε οργανώσει σεμινάρια, ειδικά στην ε, Νότια Αφρική, όπου υπάρχει ένα δίκτυο επικεφαλής ε, αποστολών, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του AIDS και έχουμε ε, προσκαλέσει και τον Γενικό Διευθυντή που βρίσκεται στην Αφρική από το Παγκόσμιο Ταμείο. Σε σχέση τώρα με αυτά που είπε ο Μισελ, το Παγκόσμιο Ταμείο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το θεωρήσει ως κάτι δικό της. Οπότε, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ή να, με κάτι να συμβάλλουμε, αυτό το κάνουμε μέσω των δικών μας ε, θεσμικών οργάνων. Γιατί, όπως είπαμε, εκπροσωπούμε πάνω από το 50% και η Κομισιόν αυτό το παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη της παρακολουθούμε και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι το Παγκόσμιο Ταμείο εξελίσσεται σε έναν τομέα και προς μια κατεύθυνση που απομακρύνεται από ε, παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο μόνο τα προγράμματα ε, και κινείται προς μια προσέγγιση πιο ενισχυτική ως προς τις ε, γενικότερες πολιτικές για την υγεία. Οπότε και με την ε, δική σας ε, συμβολή μπορέσαμε να πιέσουμε ώστε αυτό όλο να ενταχθεί στα πλαίσια του Συμβουλίου. Είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι που η πρώτη πρόταση για να υποστηριχθούν οι εθνικές στρατηγικές έχει, έχει τεθεί υπόψη του Συμβουλίου και επίσης ενισχύουμε όλες τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική του Ταμείου, οι οποίες θα το καταστήσουν πιο κεντρογενές, πιο streamlined και που θα του επιτρέψουν οι απαντήσεις που δίνουμε και οι πολιτικές που ακολουθούμε να ανταποκρίνονται στις ε, πραγματικές ανάγκες των χωρών που εμπλέκονται. Οπότε νομίζω ότι προ όφελό μα είναι και στα πλαίσια τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτέ τι δραστηριότητε του Παγκοσμίου Ταμείου, σεβόμενοι πάντα τι ιδρυτικέ αρχέ του Ταμείου. Να είναι δηλαδή πιο προσαρμόσιμο, πιο ελαστικό σε ό,τι αφορά τι ανάγκε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο συντονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση των συστημάτων υγεία. Στον τομέα λοιπόν αυτό, ενθαρρύνουμε το Παγκόσμιο Ταμείο να συμμετέχει πλήρως στις διάφορες ε, συμπράξεις που γίνονται. Και προσπαθούμε να έχουμε λίγο πιο στοχοθετημένο συντονισμό και σε ό,τι αφορά τους δωρητές για, το, για τα παγκόσμια σύστημα υγείας. Τώρα, στο Βιετνάμ, πριν από δύο χρόνια, υπήρξαν 400 αποστολές υγείας Στη Ρουάντα η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει 600, 600 ε, άτομα τα οποία ε, βρέθηκαν εκεί λόγω των, λόγω, μετά από αίτημα. Και βεβαίως εμείς παρακολουθούμε τα δραστηριότητε αυτές του Παγκοσμίου Ταμείου. Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, όπως ε, υπόθηκε, βρισκόμαστε στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος της ε, ενίσχυσης του Παγκοσμίου Ταμείου και βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των ε, ευθυνών της. Και θέλουμε στα πλαίσια αυτά να παρακολουθήσουμε και να ενισχύσουμε οικονομικά την εξέλιξη του Παγκοσμίου Ταμείου, σεβόμενοι πάντα τις αρχές χρηματοδότησης και ελπίζω να μπορέσουμε να τις προσαρμόσουμε ώστε να μπορέσουμε πιο στρατηγικά να απαντήσουμε στις αυξανόμενες ανάγκες. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Γκέρεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το θέμα που συζητούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως ε, εν ώψη των μεγάλων αποφάσεων που θα ληφθούν ε, για τη χρηματοδότηση όχι μόνο των συστημάτων υγείας, αλλά και για ε, την κλιματική αλλαγή, γιατί γενικά λαμβάνει η χώρα αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή και το θέμα είναι να μην διαφωνούμε, αλλά να θέσουμε όλα τα στοιχεία επιτάπητος και να δούμε τι χρειάζεται ο καθένας. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέμα που στέθηκε, για τον θα έχουμε εγκάρσια προσέγγιση δηλαδή, έναντι των ε, βασικών υγειονομικών συστημάτων. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Το Παγκόσμιο Ταμείο έχει προβάλει τις δράσεις, μας έθεσε σε μια θέση, σε μια θέση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τις οικονομίες κλίμακας και θα ήθελα να υπενθυμίσω το ότι το να βλέπουμε και τι έχει γίνει. Ουσιαστικά τελικά έχουμε δικαιωθεί έναντι αυτών ε, που πριν 10 χρόνια μας έλεγαν ε, ότι πρώτα πρέπει να υπάρχει πρόληψη γιατί η θεραπεία είναι πολύ ακριβή. Τελικά αυτή η προσέγγιση ήταν η κακή γιατί τα γεγονότα απέδειξαν το αντίθετο. Γιατί ποιο ε, θα είχε το κουράγιο να πάει να κάνει κάποιου ελέγχου, κάποια check-up χωρί ε, να υπάρχει ελπίδα θεραπεία. Και πριν ε, κάποια χρόνια αυτό το εκτιμούμενο κόστο που αναφερόταν τελικά δεν ισχύει σήμερα γιατί εγώ νομίζω ότι τώρα έχουμε το κόστο 150 ευρώ για έναν ασθενή στη Ρουάντα. Έτσι λοιπόν ε, διαιρέθηκε το κόστος αυτό. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι πάντοτε μας ξεπερνάει η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν πρέπει να λαμβάνουμε πιο θαραλές θέσεις και όσοι ε, είχαν το θάρρος ε, δικαιώθηκαν. Είναι πραγματικά μια ιστορία επιτυχίας. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Και θα πρόσθετα ότι χρειάζεται μια παγκόσμια προσέγγιση, μια καθολική προσέγγιση. Θα πρέπει να γίνεται το έργο σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Η Κομισιόν είχε μια προσέγγιση την οποία τη χαιρετίζω. Ήθελα να σε υποστηρίξω στην ολιστική σας προσέγγιση στον τομέα αυτό. Το θέμα είναι να δούμε πού ήμασταν πλέον επιτυχείς. Δηλαδή, αν ε, δεν είχατε γιατρούς επιτόπου, αν δεν είχατε νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να έχετε δημιουργήσει κάποιες ελπίδες για τη θεραπεία. Αυτό λοιπόν ε, συζητάμε, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη στα πλαίσια της πολιτικής ε, για την αναπτυξιακή συνεργασία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και τα προγράμματα που τέθηκαν σε εφαρμογή για την ιδρύση των νοσοκομείων, για τη συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων, μεταξύ Βορρά και Νότου, λόγου χάρη. Εγώ θεωρώ ότι στην προσέγγιση αυτή τα νοσοκομεία έγιναν κεντρικός πρωταγωνιστής ε, στην ε, ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν ε, μπορούσαμε να αναπτύξουμε τις τοπικές ικανότητες Όλα λοιπόν συνηγορούν προς τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής. Η μόνη επίπληξη που θα μπορούσαμε να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο είναι ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κονδύλια για να τα καταφέρουμε και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Κάτι τελευταίο. κατά κάποιο τρόπο το Ταμείο είναι ένα ατύχημα της ιστορίας γιατί τότε ο Μπούς δεν ήθελε να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω, δεν αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν ε, δημιουργήθηκε το Ταμείο όμως ε, τελικά μας οδήγησε σε μια τεράστια επιτυχία και πραγματικά συγχαίρω τους ηθήνοντες για το Ταμείο που πραγματικά μπόρεσαν να πετύχουν και να ε, αναπτύξουν μια τόσο καλή συνεργασία και με τα υφιστάμενα συστήματα. Πιστεύω ότι λοιπόν όλοι εδώ σε αυτόν τον οίκο σας στηρίζουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Δεκάισαρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου δεν θα είναι τόσο διαφορετική από του κυρίου Γκέρενς, ε, απλώς ε, θα το προσεγγίσω από διαφορετική οπτική γωνία. Νομίζω όπως και εκείνος ότι η λύση στο ψεύτικο αυτό ερώτημα ε, δεν είναι σε καμία περίπτωση η αμφισβήτηση του, της εγκάρσιας προσέγγισης σε σχέση με των βασικών συστημάτων υγείας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εγκάρσια προσέγγιση ενδεχομένως να είναι πιο ελκυστική για το ευρύ κοινό, γιατί ακριβώς κάνει εντύπωση, γιατί καταλαβαίνει κανείς πού πηγαίνουν τα χρήματα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ασφάλεια. Επίσης λέμε, α ναι βέβαια μπορούμε να καταπολεμήσουμε και την ελονοσία και το AIDS. Είναι κάτι που είναι πιο εύκολο να το πουλήσουμε, ας μου με πάση μου επιτραπεί η έκφραση, στον Ευρωπαίο πολίτη από ότι τα βασικά συστήματα υγεία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα όμω να επιμείνω σε αυτό που είπε ο Μισελ Ε, το ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι Μισελ. Μην πείτε σε Βελγίδα ότι δεν υπάρχουν άλλοι Μισελ, για όνομα του Θεού. 37% μας είπατε των δαπανών ε, σε μία οριζόντια προσέγγιση. Καλό είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στον ε, χαρακτήρα το περιορισμένο της γκάρσιας προσέγγισης. Αν δεν έχουμε το βασικό σύστημα υγείας, περιοριζόμαστε από ένα σημείο και μετά. Είπαμε για παράδειγμα καλό πράγμα η θεραπεία, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φαρμακεία και νοσοκομεία, όπου να μπορεί κανείς να πάρει τα φάρμακα, να υπάρξει κάποιος έλεγχος της θεραπείας κλπ. Χρειάζονται δηλαδή υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης. Με ενδιαφέρει όμως και το ζήτημα της ε, αμοιβαία ανάληψης κινδύνων στην Αφρική επειδή δεν υπάρχουν εκεί συστήματα υγείας ε, επαρκή, πώς θέλετε να πάει ο κόσμος ε, να κάνει εισφορές ή τέλος πάντων να συμμετέχει στους μηχανισμούς αλληλεγγύης, αν δεν υπάρχει δίπλα του ένα νοσοκομείο να μπορεί να πάει, ένα φαρμακείο να πάει να πάρει τα φάρμακά του ή εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο να κάνει μία εισφορά σε ένα ταμείο για κάτι για το οποίο, στο οποίο ποτέ δεν θα έχει δικαίωμα τελικά. Δίκιο έχετε κυρία Βέμπερ ότι δεν, ότι πρέπει να δούμε και τα μικρότερα προβλήματα που μπορεί να έχουν ε, σοβαρά αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διάρρεια. Μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα όπως και η ελαινοσία και η φυματίωση για παράδειγμα. Υπάρχουν όμως ε, κάποια όρια αν δεν έχουμε ένα σύστημα υγείας βασικό, ε, ένα σύστημα το οποίο δεν το έχουν αναλάβει τα ίδια τα κρατημέλη και συνεπώς δεν θα υπάρχει και πραγματική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα έχω ένα ερώτημα. Λέτε για τις στρατηγικές ε, της ε, ιατρικής περίθαλψης. Ε, μιλάμε για τα εθνικά συστήματα. Λογικό είναι αυτό. Τα κράτη-μέλη το αναλαμβάνουν αυτό. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για το εξής. Πάντοτε είχα την εντύπωση όταν πήγα για παράδειγμα στους γιατρούς χωρίς σύνορα στην Αφρική, είχα την εντύπωση πολύ συχνά ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες έτσι, συγκεντρωτικές ε, προσπάθειες ε, για το σύστημα υγείας, ε, κάτι καταπληκτικά και πολύ φανταστικά νοσοκομεία για παράδειγμα, όμως δεν γίνεται καμία προσπάθεια να κατανεμηθούν κάπως αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε α πούμε περισσότερα νοσοκομεία πιο απλά αλλά περισσότερα. Δηλαδή πρέπει να παραμείνει στα χέρια των ε, κρατών αλλά οι κυβερνήσει μερικέ φορέ έχουν πολύ μικρή τάση αποκέντρωση και συνεπώς καταστρέφουν αυτήν την ιδέα την οριζόντια. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη στους ομιλητές που δεν ήμουν εδώ από την αρχή. Αλλά, ε, κάποιες σημειώσεις από αυτά που έχασα τις ε, πήρα. Χαίρομαι για, τις, ε, για τα όσα είπε η Κομισιόν το γεγονός ότι δεν έχουμε ε, χρήματα και πρέπει να πάρουμε χρήματα και ότι το αναγνωρίζουμε είναι να βρούμε χρήματα είναι καλό. Νομίζω ότι είναι μια κοινή μας επιτυχία. Πάντα όμως θα ήθελα να σας, θα ήθελα να σας ε, ευστήσω την προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη αξία με, λιγότερη, με λιγότερες δαπάνες. Αυτό σημαίνει να, πάρουν, να, έχουμε, να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Αλλά έχουμε και του ε, στόχου τη χιλιετία για την υγεία, τα φάρμακα και πρέπει για να γίνει αυτό να υπάρξουν μακροχρόνιε ε, επενδύσει. Γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε καμία αξία για τα χρήματά μα. Ούτε θα έχουμε καμιά ιδιαίτερη, κανένα ιδιαίτερο επίτευγμα. Και σε σχέση με κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ε, ΠΟΗ αν η υποστήριξη του προπολογισμού ισχύει, τότε οι εθνικέ κυβερνήσει θα πρέπει να έχουν δυνατότητε. Δυνατότητες για τα δικά του τα προγράμματα και δυνατότητε να εκπονήσουν τι στρατηγικές του και να τι εφαρμόσουν. Με τη δημοσιονομική υποστήριξη και του, και του ownership της, ε, του επιτεύγματο που αναμένουμε, το οποίο δεν έχει μπει όμω ακόμα στην εξίσωση. Σε σχέση τώρα με την Ποτσουάνα, ήμουν επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Δύο από τους συναδέλφους μου ήταν, ε, είναι παρόντες σήμερα που ήταν στην αντιπροσωπεία και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση του θέματος του HIV και του AIDS και εντυπωσιάστηκα από το ότι ένα τρίτο του προπολογισμού πάει στην εκπαίδευση, απίστευτο, και άλλο ένα τρίτο πάει στην παροχή του 85% στην προσφορά αυτών που τον, του 85% αυτών που το χρειάζονται ε, με αντιρετροϊκά φάρμακα. Η Ρουάντα κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την ε, ε, αύξηση της ευαισθητοποίησης, γιατί αυτό ακριβώς έχει να κάνει και με την αυτοδιάθεση του καθενός που μπορεί να ε, τον εμποδίσει να καταλήξει σε μια κατάσταση που μπορεί όντω να έρθει σε επαφή με ε, μεταδοτικές ή μη ασθένειε. Έχω ένα ερώτημα τώρα για την ε, συνάδελφο από το Παγκόσμιο Ταμείο. Το 2010 είναι έτος κλειδί και σε ό,τι αφορά την επίτευξη της, παγκόσμια, της συνολικής ε, πρόσβασης σε αντιρετροϊκά φάρμακα που, για, για άτομα που έχουν HIV ή AIDS αλλά όπως είπε η Κομισιόν είναι και ο στόχος που έχουμε χρονικός χρονικός ε, για να επιτύχουμε τους ε, στόχους της χιλιετίας μέχρι το 2015. Το Παγκόσμιο Ταμείο τι ρόλο θα παίξει για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και το Παγκόσμιο Ταμείο πώς βοηθά να ε, επιτευχθούν οι στόχοι, η πρόοδος των οποίων ήταν πολύ αργή. Εντάξει, δεν είναι καλό να, βάζουμε, να κάνουμε συγκρίσει, αλλά για κάποιου στόχου, α πούμε τον 4 και τον 5, υπήρξε πάρα πολύ αργή η πρόοδο ό,τι αφορά την υγεία των μητέρων και των ε, μωρών, των παιδιών. Και αυτοί οι στόχοι τη χιλιετία πραγματικά έχουν θεωρηθεί προτεραιότητα και από το ΟΗΕ και από την Καναδική Προεδρία του G8. Οπότε πραγματικά θα ήθελα την απάντηση στην ερώτησή μου αυτή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τις συμβολές του σήμερα το πρωί και τις παρατηρήσεις τους και τον ΑΠΟΗ και την Κομισιόν και το Παγκόσμιο Ταμείο. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να επιτύχουμε τους ίδιους στόχους, οπότε μόνο μέσω της συνεργασίας και της ε, έβρεσης των ε, κενών που υπάρχουν και των ελλείψεών μας, μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μέχρι τις 5 η ώρα και έχουν ζητήσει ακόμη τέσσερις συνάδελφοι το λόγο. Θα θέσουν τις ερωτήσεις και κατόπιν θα πρέπει να ξαναδώσουμε το λόγο στους ομιλητές. Έτσι λοιπόν θα σας ζητούσα να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Ο κύριος Δέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στην αρχή της συζήτηση. Θα πρέπει να παραβρεθώ στην ε, Επιτροπή για τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα και στην Επιτροπή ε, που συζητά τα θέματα Βορρά Νότου. Δύσκολο λοιπόν να είμαι παντού. Αναγνωρίζω τη μεγάλη επιτυχία του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση της ελληνοσίας, του AIDS και της φυματίωσης. Παρακολουθώ το έργο του πολύ κοντά και θα ήθελα να ρωτήσω τα δύο εξής. Πιστεύετε ότι τώρα έχουμε συγκρατήσει μία ενδυνάμει επιδημία και μπορούμε να περιμένουμε να μειωθούν τα νούμερα σε όλες τις χώρες πέραν της Ινδίας. Και δεύτερον, Υπάρχει και άλλη μια νόσος ε, η οποία κάθε χρόνο σκοτώνει 5 εκατομμύρια παιδιά και μιλάμε για τις ε, ασθενείες που πλήττουν τα παιδιά όπως η διάρρεια ε, και αυτές σκοτώνουν περισσότερα παιδιά από τη λονοσία και η φυματίωση μαζί. Γιατί δεν ενδιαφέρεται κανείς για μια ασθένεια που σκοτώνει 5 εκατομμύρια παιδιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μου δίνετε πάντα το λόγο αφού κάνετε την προειδοποίηση να είμαστε σύντομοι, έτσι θα υποβάλω μόνο τις ερωτήσεις μου, παρόλο που θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή. Έχω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Καζατσκίνε, αν το λέω σωστά. Πώς ξεπερνάτε τα προβλήματα κυβερνητικής διαφθοράς και της διαφθοράς της εξουσίας, δεδομένου ότι μας έχετε πει ότι έχετε κάνει πάρα πολλά προς την κατεύθυνση αυτή στις χώρες που χρειάζονται. Και δεύτερο, μας έχετε μιλήσει για το σημαντικό ρόλο των ευρωβουλευτών και των βουλευτών στην στήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου και θα ήθελα να γίνετε πιο σαφείς, να μας πείτε τι ακριβώς περιμένετε από μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχω και δύο ερωτήσεις προς την κυρία Βέπερ. Η πρώτη ερώτηση αφορά το γεγονός ότι δεν χορηγούνται φάρμακα για το AIDS, αντιϊκά φάρμακα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε μια περιοχή αναλυτής που να επιβεβαιώνει εργαστηριακά ότι το άτομο πάσχει πραγματικά από AIDS. Καταλαβαίνετε ότι αυτό καταδικάζει εκατομμύρια ανθρώπους ενώ γνωρίζουμε κλινικά περίπου ότι πάσχουν από AIDS να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα. Και ο κάθε αναλυτής κοστίζει μόνο 15.000 δολάρια. Θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να εγκατασταθούν σε περιφερειακό επίπεδο αυτοί οι αναλυτές ούτως ώστε να μην στερούμε ενώ υπάρχουν φάρμακα για το AIDS να, να μην στερούνται αυτά τα άτομα της ε, θεραπείας. Και δεύτερο, κυρία Βέμπερ, έχετε κάποιο πρόγραμμα για την λωρίδα της Γάζας, μιας περιοχής που βρίσκεται μόνο 20 λεπτά μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό, δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα και μόλις ο πληθυσμός, ζουν 2 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι εκεί μέσα, μόλις ο πληθυσμός καταφέρει να φτιάξει ένα υποτυπώδες σύστημα αποχέτευσης, έρχονται κάποιοι και το βομβαρδίζουν και το καταστρέφουν. Δηλαδή, ποια πολιτική παρέμβαση γίνεται προ την κατεύθυνση του Ισραήλ για να εξασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στοιχειοδό παροχή τρεχούμενου νερού και αποχετεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. La parole est à Madame Keller. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση που δεν αφορά αμέσως τα βασικά συστήματα ή τα εγκάρσια ταμεία, αλλά έχει να κάνει με τα κονδύλια που αναφέρθηκαν και καθώς εδώ έχουμε εμπειρογνώμονες που εργάζονται ε, στα θέματα ανάπτυξης και υγείας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε η συμφωνία ΑΚΤΑ πώς θα επιδράσει στην πρόσβαση στα φθηνά φάρμακα καθώς ε, ξέρουμε ότι τα φάρμακα που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι πάρα πολύ ακριβά και η πρόσβαση στα γεννόσιμα φάρμακα είναι πιο εύκολη και καλό και σύμφωνα με την ΑΚΤΑ ε, προβλέπεται ότι θα πρέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να ισχύουν ε, και για τις χώρες διέλευσης όχι μόνο εμπορίας. Θα ήθελα λοιπόν να πείτε πώς θεωρείτε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των θεμάτων αυτών. Ναι, θα μιλήσω πολύ λιγότερο από δύο, από δύο λεπτά. Υπάρχει μια σειρά νόσων στον κόσμο που μας ανησυχούν πάρα πολύ κυρίως ε, γιατί αφαιρούν τη ζωή εκατομμυρίων ε, ατόμων και αναφερόμαστε εδώ στο AIDS, στη φυματίωση, στην ελονοσία κτλ αλλά πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες αυτές. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να ξεχάσουμε ότι τα συστήματα υγείας είναι δομές, γενικές δομές που ε, χρησιμεύουν στον πληθυσμό από μια σκοπιά πρόληψης αλλά και μια σκοπιά θεραπείας και όσο διατηρούμε την προσπάθεια για να εξαλείψουμε ορισμένε νόσους, θα πρέπει ταυτόχρονα να εστιάσουμε και στο να υποστηρίξουμε τα δημόσια συστήματα υγείας και τους μηχανισμούς πρόσβασης όλων των πολιτών με ισότιμο τρόπο σε αυτά τα συστήματα υγείας. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή η αρχιτεκτονική της βοήθειας και της στρατηγικής της επικοινωνίας για τον τομέα της υγείας που προετοιμάζει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις στρατηγικές των χωρών δικαιούχων. Αναφέρομαι στις γενικές στρατηγικές για την καταπολέμηση των ασθενών αυτών και για την φροντίδα της υγείας των πολιτών. Δεν θα ήθελα να αναφέρεστε μόνο σε πολύ συγκεκριμένες ε, νόσους. Θα πρέπει να ε, φροντίζουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε επαρκή στήριξη για να κατεπολεμήσουμε και τις νόσους που αφαιρούν εκατομμύρια ζωές. Μάλιστα τώρα ε, ο κάθε ομιλητή έχει πέντε λεπτά για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Καταρχήν ο κύριος Κατσάτκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω πολύ σύντομα με τις, στις πολλές ερωτήσεις που μου ετέθησαν, αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε τέσσερις από αυτές και αντιστοιχούν σε τέσσερα ζητήματα. Καταρχά, αυτό το θέμα των συστημάτων υγείας. Ευχαριστώ πολύ όσους πήραν το λόγο, γιατί είπαν ότι δεν πρόκειται να φέρουμε σε ανταγωνισμό το οριζόντιο με το εγκάρσιο. Θέλουμε απλώς να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος ε, που, που μας οδηγούν στο να πούμε ότι ε, θα πάμε προς, την κατεύθυνση των συστημάτων υγείας και μετά η υγεία κάποια στιγμή θα επέλθει και αυτό θα μας ανταμείψει. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, βέβαια να παραγνωρίσει κανείς την ελονοσία, την ελονοσία, τη φυματίωση ή το AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα συστήματα υγείας και οι ασθένειες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα πλήρες πλαίσιο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και αναφέρθηκα προηγουμένως σε ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Αιθιοπία χρησιμοποίησε τα ε, ταμεία για το AIDS και για την ελονοσία για να υπάρξουν σταθμοί περίθαλψης, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων περίθαλψης που όχι μόνο δίνουν αντιρετροϊκά φάρμακα ή ε, εκπαιδεύουν ε, το κόσμο στο πώς να χρησιμοποιεί τις κουνουπιέρες για παράδειγμα, αλλά τους ενημερώνουν και για την αναπαραγωγική υγεία ε, και για τις διάφορες θεραπείες, για τις έντονες οξύες λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα τις διαρροικές ασθένειες των παιδιών. Γνωρίζω ότι το AIDS και τέτοιου είδους ασθένειες τυχαίνουν πάντοτε μεγάλη προσοχή 45% των γυναικών από 15 έως 50 ετών στην Αφρική πεθαίνουν από AIDS και ένα, ένας ακόμη τρόπος ε, να τις βοηθήσουμε είναι να τις απελευθερώσουμε από τη μάστιγα αυτή. Η εκπρόσωπο στη Ρουάντα, στη Γενέβη, μας είπε ότι μέχρι πριν από τέσσερα ε, πριν από τέσσερα χρόνια τα παιδιά ήταν δύο-δύο στα κρεβάτια των νοσοκομείων για τέτοιες βασικές ασθένειες ε, και μετά, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια μπορούν πια τα νοσοκομεία να θεωρούνται πράγματι νοσοκομεία ε, της, δηλαδή με την έννοια της πραγματικής ε, παροχής περίθαλψης. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας πώς θα καταφέρουμε και συγγνώμη κιόλα που τα λέω έτσι λίγο γραφικά. Ένας υπουργό Υγείας ε, με φοβερές ιδέες για, το, για την ε, μεταρρύθμιση της, ε, του στήματος υγείας της χώρας του. Όμως, εμείς τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι μόνο από τον Υπουργό Υγείας. Αντιθέτως, υπάρχει ο μηχανισμός συντονισμού της χώρας στον οποίο εκπροσωπούνται η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, αλλά και το Υπουργείο Γυναικών, το Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως ε, και η κοινωνία των πολιτών. 40% μάλιστα συμμετοχή έχει η κοινωνία των πολιτών Όσοι έχουν λοιπόν ε, ε, προσβληθεί από τις ασθένειες, οι συνάδελφοι από τη UNICEF ε, ή του προγράμματος για το AIDS, όπως είπε η συνάδελφος προηγουμένως, όλοι μαζί επεξεργάζονται τις προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση που θα ζητήσει μια χώρα από το Διεθνές Ταμείο. Για τα δύο ερατήματα σχετικά με το ποιες είναι οι ελπίδες μας σε σχέση με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Είναι γεγονός ότι με την ελονοσία η κατάσταση είναι δύσκολη. Νομίζω ότι πριν από το 2015 θα επιτύχουμε όμως τους σχετικούς ε, στόχους ε, της χιλιετίας και νομίζω ότι καλά τα πηγαίνουμε και στην περίπτωση της φυματίωσης ε, με την εξαίρεση βέβαια της απειλής της αύξησης της ανθεκτικής φυματίωσης. Ως προς το AIDS ελπίζουμε ότι θα εξαλείξουμε σχεδόν ε, την μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο παιδί και να σώσουμε εκατομμύρια άλλες ζωές με την πρόσβαση στη θεραπεία. Ναι, έχουμε καθυστερήσει στον αναπτυξιακό στόχο 5, ειδικότερα όσον αφορά την ε, μητρική θνησιμότητα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Αλλά σας το είχα πει, σας το είπα ε, κυρίες και κύριοι, αν δεν υπάρχουν πόροι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Απλά είναι τα πράγματα και γι' αυτό πιστεύω ότι το ζήτημα που τίθεται στο 2010, όταν βλέπει ο κόσμος ε, την ε, καθυστέρηση για το στόχο 5, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους που πρέπει να αφιερωθούν ε, στην μητρική θνησιμότητα και στη συνέχεια υπάρχει μια ολόκληρη εθνική συζήτηση κατά πόσο το Διεθνές Ταμείο πρέπει να είναι ο μηχανισμός, ο φορέας αυτών των κονδυλίων προς τη χώρα. Όσον αφορά τη διαφθορά τώρα, Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αναφέρω λεπτομερώς όλους τους μηχανισμούς ε, που έχουμε ε, στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι το Διεθνές Ταμείο ανταποκρίθηκε στην διεθνή κοινότητα δείχνοντας ότι επαγρυπνεί πραγματικά σε σχέση με, την, ε, με το πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια. Είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις, τους λάθος συναγερμούς Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς αυτό και παρά τις διάφορες προειδοποιήσεις. Ε, αν πάτε στον ιστότοπό μας ε, θα δείτε όλες τις εκθέσεις των επιθεωρητών μας. Όλα αναφέρονται εκεί για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες χώρες προσπάθησαν ε, με λάθος τρόπο να χρησιμοποιήσουν κάποια κονδύλια ή μέτρα που είχαμε λάβει. Όσον αφορά το, τους ρόλους του Κοινοβουλίου. Τέσσερις. Πρώτον, να συμμετέχουμε στην έκκληση για την υγεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης διακόπτη πρόεδρος. Παρακαλώ, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει επίσης να ενημερώσουμε, συνεχίζει ο μιλητής, ε, την, ε, τους πολίτες ε, και επίσης να ενημερώσετε, τους, να υποστηρίξετε τους συναδέλφους σας από τον Νότο για να μπορέσουν και εκείνοι να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρηση. κυρία Βέμπερ Μένστορφ. Ο πιο σημαντικός στόχος είναι η πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίες υγείας, σε φτηνές, σε φτηνά ε, φάρμακα, τα κράτη-μέλη της ΠΟΗ έχουν διαπραγματευτεί μια νέα στρατηγική για την κοινοτομία, για τη δημοσία υγεία, ώστε να συγχωνευτούν όλες αυτές οι διαφορετικές πτυχές μεταξύ των δικαιωμάτων και των εμποδίων που υπάρχουν για να επιτευχθεί ο στόχος των φτηνών φαρμάκων. Εκεί όντω υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκή πολιτική να ε, δεχτούμε τις, ε, την ε, ευελιξία του τρίψ και να προσπαθήσουμε να βρούμε πώς θα προωθηθούν οι πολιτικές. Ε, η παγκόσμια πρόσβαση πρέπει να αφορά χώρες και όπως η Αφρική. Γιατί εκεί οι φτωχοί από το ειστέρημά τους προσπαθούσαν να ενισχύσουν τις υπηρεσίες υγείας. Οπότε υπάρχει περιθώριο για κοινωνική προστασία. Η κοινωνική προστασία είναι πολύ σημαντική και αυτή είναι μια πρωτοβουλία που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί λοιπόν πρέπει να πιέσουμε, να προστατεύσουμε τους πολίτες, να τους δώσουμε μια αλφα ασφάλεια για το μέλλον. Έχουμε την εμπειρία εδώ στην Ευρώπη. Με τα συστήματα υγείας και τι γίνεται όταν οι κυβερνήσεις προωθούν μόνο τα νοσοκομεία. Νομίζω εδώ πρέπει να παίξουν ρόλο τα εθνικά προγράμματα υγείας και οι εθνικές πολιτικές, να δούμε δηλαδή ποιε είναι οι ανάγκε να τι αξιολογήσουμε και να μιλήσουμε και για προτεραιότητες. Αυτό που πρέπει να γίνει από κοινού με την πρωτογενή ε, υγειονομική περίθαλψη είναι να προστατεύσουμε τις κοινότητε να δώσουμε ε, υπηρεσίες υγείας στους ε, πολίτε. Αυτό είπε και ο εκπρόσωπος λίγο πιο πριν. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αιτίε. Ας πούμε, το πρόβλημα της διάρειας. Στην Ινδία όμως υπάρχει και άλλη επιδημία του διαβήτη. Τα συστήματα υγείας λοιπόν πρέπει να λάβουν υπόψη τους στις στρατηγικές τους αυτές τις ασθένειες και να φαίνεται αυτό, να φαίνεται δηλαδή πώς μπορούν να δοθούν τα φτηνά φάρμακα σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Γάζα, η ΠΟΗ προσπαθεί να ενισχύσει τις εθνικές στρατηγικές, γιατί όντω το θέμα της αποχέτευσης και του νερού είναι πραγματικά σημαντικό. Για τη χρηματοδότηση, κάτι που ξέχασα, νομίζω ότι οι δωρητές στο Παγκόσμιο Ταμείο θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε αυτές τις ακριβώς τις ασθένειες. Και σε ό,τι αφορά τη γενικότερη διακυβέρνηση, είναι σημαντικό όχι απλώς να είμαστε συνεκτικοί στην παροχή υπηρεσιών, αλλά να είμαστε συνεκτικοί και σε ό,τι αφορά τι πολιτικές μας, πολιτικές υγεία. Και να είμαστε συνεκτικοί σε ό,τι αφορά και τι εντολέ που δίνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριάρα έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι μάλλον δεν έχετε χρόνο. Και καθώς εγώ θεωρώ ότι και εγώ ανήκω εδώ στον Νίκο, θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω όλους όσους εξέφρασαν την ε, υποστήριξή τους ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πώς προσεγγίζει το θέμα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι η ανακοίνωσή μας για την παγκόσμια υγεία θα μας δώσει ευρείες ευκαιρίες να κάνουμε μια συζήτηση εις βάθος, όπως ε, υπόθηκε και από τον κύριο Κάτσμαν. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε στην ίδια βάρκα και κοπηλατούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Και ε, θεωρώ ε, ότι όσα θα σας παρουσιάσει και ο κύριος Πίμπαλξ τις επόμενες εβδομάδες ε, θα σας δώσουν και σε εσάς και σε εμάς την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στη συζήτηση. Ε, πραγματικά είμαστε σε μια πολύ σημαντική χρονιά. Έχουμε τη συνδιάσκεψη για τους στόχους της Λετίας στη Νέα Υόρκη, την αναστήσεως των ταμείων. Συζητούμε το θέμα της προσέγγισης της υγείας από μια συστηματική σκοπιά Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να ανταποκριθούμε και στην πρόκληση για το στόχο 5. Αν πραγματικά κάπου χρειάζεται συστημική απάντηση είναι για το στόχο της χιλιετίας υπαριθμών 5. Ελπίζω λοιπόν ότι έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τις συζητήσεις. Να αναφερθώ και στο όσα είπε η κυρία Κέλλερ Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην ανακοίνωσή μας είναι το θέμα της γνώσης, η πρόκληση της γνώσης. Και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά μπορούμε να συζητήσουμε ένα από τα βασικά θέματα έτσι, που αφορά τη διάθεση των φαρμάκων σε λογικές τιμές ε, προκειμένου να ε, είναι δυνατό η προτεραιότητα της υγείας να είναι προσβάσιμη σε όλες. Σας ευχαριστώ και εμπομονώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές σας. Τώρα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Περιμένουμε τον ε, κύριο Επίτροπο που θα παρευρεθεί εδώ για να μιλήσουμε για τις νέες προκλήσεις.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 Πάμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξή μας ε, που έχει να κάνει με την παρουσίαση και τη συζήτηση των ομάδων, της ομάδας εργαστηρίων ιδεών με τίτλο «Νέες προκλήσεις, νέα αρχή. Τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Συνεργασίας». δεν είναι μόνο πολύ επίκαιρο, είναι και αρκετά τολμηρό γιατί προτείνει μια, ένα νέο όραμα της ανάπτυξης, ένας νέο, ένα νέο τρόπο εργασίας ε, σε νέες παγκόσμιες προκλήσεις. Έχουμε παρόντες ερευνητές ε, εξέχουσες προσωπικότητες ε, στις, από τις τέσσερις οργανώσεις και θα σας πω τα ονόματα Simon Maxwell, ερευνητής στο Overseas Development Institute in London, Dirk Messner, διευθυντής ε, του Γερμανικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης στη Βόνη, Paul Engel, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναπτυξιακής Πολιτικής και Διαχείρισής της στο Μάστριχτ και Richard Youngs, διευθυντής του ΦΡΙΝΤΕ στη Μαδρίτη. Επίσης είναι παρόν ε, ο Επίτροπος Άντρης Πίμπαλξ, ε, ο οποίος δέχτηκε με χαρά την πρόσκλησή μας να παρευρεθεί στις σημερινές μας εργασίες. Ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, Επίτροπε, για την παρουσία σας. Σας είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα να δώσω ευθύ αμέσω τους εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων των εκθέσεών τους. Πρώτα, ο κύριος Μάξουελ για πέντε λεπτά. 15 λεπτά, αλλά θα τα μοιραστούμε και είμαστε τρεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική χρονική στιγμή επειδή ενισχύεται η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και η ομάδα του κυρίου Πίμπαλξ. Οπότε είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι. Έχουμε αυτή την έκθεση που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε βεβαίως να σας δώσουμε αντίτυπα και ελπίζουμε ότι σε μερικά χρόνια θα είναι πολύ πολύτιμη τρία ζητήματα στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Το πρώτο είναι τι είναι αυτό που πραγματικά μας ενθουσιάζει, δεύτερον, τι είναι σημαντικό και το τρίτο είναι τι είναι πολιτικός εφικτό υπό τις ε, συνθήκες αυτή τη στιγμή με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχουμε. Και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς και ελπίζουμε η συνεισφορά μας να είναι όσο το δυνατόν πιο θετική. Για 10 χρόνια οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας ε, έχουν επικρατήσει στις συζητήσεις μας και παραμένουν σημαντικοί, ειδικότερα το 2010, επειδή θα γίνει σύνοδος κορυφής το Σεπτέμβριο. Για όσους όμως ε, εργάζονται σε διεθνές επίπεδο κάθε μέρα, όπως εμείς, ε, οι προτεραιότητες αλλάζουν πολύ γρήγορα. Η οικονομική κρίση μας υπενθύμησε πόσο σημαντικό είναι η παγκοσμιοποίηση να λειτουργεί και για τους φτωχού, αλλά και, για τους και όπως και για τους πλούσιους πλούσιους, ε, η ε, διατροφική ε, κρίση, Είχαμε πολλά προβλήματα πέρσι και επειδή έχουμε και τη μεγάλη πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και το θέμα των ευάλωτων χωρών που θα είναι τμήμα της, του προγράμματος για την ανάπτυξη κατά τα επόμενα έτη, δεν πρέπει άλλα ζητήματα να μην τα λαμβάνουμε υπόψη, γιατί ακριβώς διαμορφώνουν την άποψή μας και την προσέγγισή μας για την υγεία, για την ε, ε, εκπαίδευση, για την ανάπτυξη. Δεν θέλουμε λοιπόν να σταματούμε να προσέχουμε τους στόχους της χιλιετίας, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε και άλλα προβλήματα που προκύπτουν και θα σας πει περισσότερο ο συνάδελφος ε, σε λίγο. Δύο βασικά πορίσματα. μία από τις δύο προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αναπτυξιακή βοήθεια και μόνο. Είναι σημαντική, αλλά είναι ένα τμήμα της ε, προσπάθειας. Ε, πρέπει να έχουμε και ε, άλλες πολιτικές και διπλωματία. χρειάζεται μια γενικότερη υποστήριξη της προσπάθειας. Επίσης, όλες αυτές, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουμε μερικές φορές ξεφεύγουν πια από τα εθνικά όρια και πηγαίνουν σε μια πολυμερή διεθνή αρένα και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ομοιάζει υπ' αυτήν την έννοια ε, με τον ΟΗΕ για παράδειγμα ή την Παγκόσμια Τράπεζα. Όταν όμως αποφασίζεται πώς, ε, πώς θα διαθέσει ε, τους πόρους της, τουλάχιστον στη δική μου χώρα, οι υπουργοί λένε θα κάνω προσπάθεια να επιλύσω προβλήματα διμερώς με τους συναδέλφους μου ή στο πλαίσιο του ΟΗΕ στην Παγκόσμια Τράπεζα ή θα συζητήσω το θέμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσω να το επιλύσω. Κοιτάξτε, η άποψή μας είναι η εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει πολλά λεφτά, πολλά λεφτά και πάρα πολλά δημόσια αγαθά, αλλά δεν έχει το, την, ε, τον πολιτικό τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπα... Ε, ο ΙΕ έχει λογοδοσία, έχει άλλα πράγματα, αλλά δεν έχει πάντοτε τα χρήματα ούτε και τις κοινέ αξίες να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει κοινέ αξίες, έχει πόρους και υπάρχει και μια ποικιλία μέσων. Το μόνο που μπορούμε, το, αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να τα συντονίσουμε. Για να δούμε τι γίνεται διεθνώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί σε συζητήσει για του ε, αναπτυξιακού στόχου ε, πριν από το Σεπτέμβρη. Προβληματισμό για τον ρόλο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο τώρα στο συντονισμό το μακροοικονομικό η Παγκόσμια Τράπεζα όλο και περισσότερο αυξάνει τις δαπάνες της και όλο και περισσότερο διαχειρίζεται τη, τα κονδύλια για την κλιματική αλλαγή ε, και θα υπάρξει μεγάλη ποικιλία μέσων προς αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς αναρωτιόμαστε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θέτει επιτάπητος, ε, ποια πόρτα θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα μπορέσει να ε, αξιοποιήσει την ευκαιρία μιας ισχυρής Επιτροπής Ανάπτυξης και μιας νέας ηγεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην είναι μόνο ένα, μια παγκόσμια ατζέντα, αλλά να είναι δική μας ατζέντα. Και πρώτα θα σας μιλήσει ο συνάδελφος ε, για περισσότερες λεπτομέρειες. Θα χρησιμοποιήσω 3-4 λεπτά για να μιλήσω για τις ε, κλιματικές αλλαγές. Το αναφέρομαι και στην έκθεσή μας, αλλά νομίζουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ε, απειλή για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Και αυτό ο τομέα πολιτική, για αυτό το τομέα πολιτική, είναι πρωτοπόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει όντω να δώσουμε κάτι, να βάλουμε κάτι επιτάπητο όταν μιλούμε για θέματα κλιματικών αλλαγών. Αν σκεφτείτε λοιπόν την πολιτική για το κλίμα, σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική, μιλούμε για συνεκτική πολιτική, γιατί πρέπει δηλαδή να συνδυάσουμε διάφορου τομεί πολιτική ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Μιλούμε για αναπτυξιακή πολιτική, δραστηριότητε στι αναπτυσσόμενε χώρε, μιλούμε για την ενεργειακή μα πολιτική στην Ευρώπη και παγκοσμίω, μιλούμε για την εξωτερική πολιτική, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τι δυνατότητε που έχουμε στα πλαίσια τη εξωτερική μα πολιτική και στα πλαίσια τη διπλωματία, ώστε να οργανώσουμε ε, ομάδες ε, πρωτοπόρων εξωτερική πολιτική και στι ε, βιομηχανοποιημένε και στι αναπτυσσόμενε χώρε. Οπότε η κλιματική αλλαγή είναι ένα τομέα όπου η Ευρώπη πραγματικά θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Τρία σημεία. Ένα. Για τη δημιουργία ενό νέου οροσίμου μετά την Κοπεχάγη. Να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, να επενδύσουμε στην εμπιστοσύνη. Γιατί μετά από την Κοπεχάγη φύγαμε χωρί να υπάρχει, με, με, έτσι με έλλειψη εμπιστοσύνη. Και μετά την Κοπενχάγη είχαμε την εντύπωση ότι η παγκόσμια κοινότητα δεν ήταν σε θέση να οργανώσει, να διαχειριστεί τέτοια μεγάλα ε, γεγονότα κοινού, συμφέροντο για να αντιμετωπίσει τι κλιματικέ αλλαγέ. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε χρήματα στι ε, διάφορε πρωτοβουλίε για τι αναπτυσσόμενε χώρε, για τι πρωτοβουλίε για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το ορόσημο στην πολιτική ζωή και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, να ε, ε, ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια επίθεση, επί, παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ε, πρόκληση σε ό,τι αφορά την νοοτροπία. Εδώ η Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει για την κλιματική αλλαγή και η αναπτυξιακή πολιτική. Έχει να κάνει με το πώς μπορούμε παγκοσμίω να, εργα... να οργανώσουμε την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τη χρήση χαμηλού άνθρακα. Και μιλούμε και για την απάλληψη της φτώχειας και την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στα πλαίσια της μείωσης, της δραστικής μείωσης και παγκοσμίω, αλλά και σε, α, όχι μόνο στις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις εκπομπές άνθρακα. Η Κοπεχάγη λοιπόν απέτυχε και επειδή πολλές, πολλοί, πολλοί πολιτικοί δεν πίστεψαν ότι αυτό μπορεί να γίνει, είναι εφικτό. Και η ανάπτυξη και η ε, ε, αντιμετώπιση της φτώχειας και η μείωση του άνθρακα δεν πίστεψαν ότι είναι εφικτό η Ευρώπη είναι ένα εργαστήριο για την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τη χρήση χαμηλού άνθρακα, ε, τη χαμηλή χρήση άνθρακα, συγγνώμη. Ε, οπότε ξέρουμε ότι στην, και στην ε, Παγκόσμια Τράπεζα και στην, ε, υπάρχουν ομάδες που μπορούν να προωθήσουν αυτές τις, προ, τις πρωτοβουλίες, αλλά εμείς ως ομάδα σκέψης είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να κάνουμε την έρευνα, υπάρχουν οι δυνατότητες ε, έρευνας που μπορούν να μεταφραστούν σε προγράμματα που να μπορούν να λειτουργήσουν επί τόπου. Δεύτερο είναι αυτό λοιπόν. Και πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιε πρωτοβουλίε για την ε, χαμηλή χρήση άνθρακα. Επίση, κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω. Η πολιτική για το κλίμα χρειάζεται ομάδε πρωτοπόρων στον παγκόσμιο χάρτη για να είναι επιτυχής το πιο εκνευριστικό στην Κοπενχάγη ήταν ότι η Ευρώπη ήταν μόνη τη όταν προσπαθούσε να προωθήσει την ε, ατζέντα για το κλίμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν εταίρου. Η αναπτυξιακή πολιτική είναι ένα κομμάτι του παζλ, ένα εργαλείο για να συνεργαστούμε ω κράτη που έχουν στόχο και έχουν δεσμευθεί να, να μειώσουν τη χρήση άνθρακα. Έτσι μπορούμε μόνο να καταλήξουμε σε ένα καλό καθεστώ για την χρήση του άνθρακα στο μέλλον. Η αναπτυξιακή πολιτική λοιπόν τώρα εδώ, από με την, με την εξωτερική πολιτική και την ενεργειακή πολιτική, μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Η πολιτική λοιπόν για το κλίμα είναι ένα χώρο, ένα τομέα όπου η πολιτική η συνοχή είναι σημαντική και εδώ η Ευρώπη έχει πραγματικά το συγκριτικό πλεονέκτημα για να προωθήσει την ε, ατζέντα. Ευχαριστώ. Εμείς από τη δική μας ε, πλευρά θα θέλαμε να αναφερθούμε στο θέμα της ε, πολιτικής συνοχής και στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Ένα θέμα που τονίστηκε και σε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θέλουμε να δούμε και τι χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσουν τα θέματα αυτά και μάλιστα στα πλαίσια της ανάπτυξης ε, δύο καθήκοντα. Νομίζω ότι το πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχει όλα τα μέσα και τώρα έχει έρθει το πληρώμα του χρόνου να βάλουμε τα χρήματα, ε, να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για τους κατάλληλους σκοπούς. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, έχουμε τον κώδικα δεντολογίας και μπορούμε να έχουμε και ένα πρόγραμμα εργασίας PCD ε, που να είναι ορθά προσανατολισμένο. Όμως, ε, ο διάβολος κρυβέται στις λεπτομέρειες και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πραγματικά μεγάλο μερίδιο ευθύνης ε, που πρέπει να αναλυφθεί μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να προωθηθούν περαιτέρω οι δεσμεύσει αυτέ. Γιατί το λέμε αυτό γιατί σε όλες ε, τις μελέτες που υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα και εμείς και οι συνάδελφοί μας, υπάρχει πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη μόνο όταν υπάρχει πολιτική βούληση και δέσμευση για να σημειωθεί πρόοδος. Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε αρκετά πράγματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και τα οποία συνάδουν με τη συζήτηση που έχετε στον οίκο αυτό. Ένα από αυτά είναι να υπάρχει από αποτελεσματική επικοινωνία με τα Εθνικά Κοινοβουλία και με την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Ε, να υπάρχει καλύτερη κατανομή της εργασίας και η πολιτική συνοχή. Αυτά συνεισφέρουν ε, το να επιτευχθούν τα συμφέροντα όλων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργηθούν συνέργειες για την ανάπτυξη και σε άλλους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ε, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το πόσο ε, δύσκολο είναι, παραδείγματος χάρη, να έχουμε μια συνολική εταιρική σχέση με την Αφρική λόγου χάρη και να αναφέρω κάτι που είναι τεχνικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενωπημένα κριτήρια για να αξιολογήσουμε την πρόοδο, να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα εργασίας PCD και να αξιολογήσουμε και το πώς λειτουργεί ο κώδικας τεχνολογίας. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ε, να έχουμε και αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεν ξέρουμε Πώ ακριβώ θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε επαρκέ προσωπικό που να έχει δεξιότητες ε, για τα θέματα της ανάπτυξης, να βλέπουμε ε, να υπάρχει δυνατότητα ή χωρίς δικαιούχοι να μας επισημάνουν που έγκυται οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής και φυσικά περιμένουμε από τον αρμόδιο επίτροπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν και τον τελικό λόγο στην ανάπτυξη των προγραμμάτων Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό των αντιπροσωπιών. Πιστεύουμε ότι οι αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Αν θέλετε να έχετε αποτελέσματα στον τομέα του κώδικα δοντολογίας, θα πρέπει να ξεκινήσετε ένα διάλογο με τους εταίρους επιτόπου σε επίπεδο χωρών. Και επίσης θα πρέπει να παρουσιαστούν ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα επί των προτάσεων που έχουν υλοποιηθεί. λόγω χάρη να υπάρχει λογοδοσία ε, για την εφαρμογή των πολιτικών ε, δέσμευση PCD στις πολιτικές ομάδες και στις επιτροπές. Θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να γίνονται μελέτες αντικτύπου για μη αναπτυξιακές πολιτικές και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό προσπαθείς ε, να εμπλακεί περισσότερο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Ευχαριστώ. Um, Κάτι ακόμη που εξετάζουμε στην έκθεσή μας ε, είναι οι ευάλωτες χώρες, η αναπτυξιακή πολιτική εκεί. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο σε σχέση με τη σύνδεση της ασφάλειας και, την σύνδεση, και την, της ανάπτυξης συγγνώμη, και πιστεύουμε ότι σε αυτό το τομέα μπορεί να σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκρεμείς ε, συγκρούσεις, ε, οι συγκρούσεις που δεν έχουν ε, σταματήσει, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν κάποιες αιστείες και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της, πολιτική, της πολιτικής μας είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα να πρωτοστατήσει επειδή έχει μεγάλη εμβέλεια μέσων πολιτικής. Υπήρξαν αυξήσεις αναπτυξιακή συνεργασίας από τους Ευρωπαίους δωρητές προς τις ευάλωτες χώρες, αλλά ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μερικές περιπτώσεις ακόμη όπου υπάρχουν ε, πιθανότητες ε, ανάπτυξης συγκρούσεων όπου δεν επενδύει επαρκώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, Πακιστάν, Ιράκ, Νιγηρία, Σουδάν, Σομαλία. Και ένα γεγονό που μπορεί να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι το Πακιστάν ε, δεν λαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια ή λαμβάνει λιγότερη από άλλες ε, χώρες που βρίσκονται στην Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Όλες, όλοι αυτοί οι λόγοι για υπέρ της ε, ε, μεγαλύτερης ασφάλειας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη δεν έχουν μεταφραστεί στην πράξη σε τίποτα. Δεν ε, είχε ως αποτέλεσμα τόσο μακροχρόνια ανάπτυξη γιατί ακριβώς ε, δεν υπήρξε καλή διαχείριση των ε, κρίσεων. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών μέσων ε, για, σε περίπτωση συγκρούσεων, για παράδειγμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη αγωνίζεται να περάσει από τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση κρίσεων σε μια πιο μακροπρόθεση συμμετοχή ε, αντιμετώπισης των ε, αιτίων ε, της των συγκρούσεων. Έχουμε 24 αποστολές, αλλά δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να ε, άρουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν για την ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες που πηγαίνουν εκεί επί τόπου και ακόμη δεν έχουν με απτό τρόπο επηρεάσει τα πράγματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, έχει πράγματι αναπτύξει ε, μέσα ανάπτυξη στις χώρες αυτές ε, και ειδικότερα στις χώρες όπου υπάρχει αρκετή ανασφάλεια ε, και συνεπώς υπάρχει και κάποιος κατακαιρματισμός ε, των αναπτυξιακών πόρων. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Αφρικανική Ένωση, πρέπει να υπάρξει και κάποια πολιτική όθηση και αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Κάτι ακόμη, 25 πυρογνώμονες από τέσσερα think tanks ε, και αν νομίζετε ότι 25, μέλη του κοινοβου... 25 χώρες μέλη είναι δύσκολο να, να, να αποφασίσουν κάτι, φανταστείτε τι, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα κάποιος είπε, ε, το... ότι... κάποιος είπε ότι αν ας πούμε μεταξύ των οικονομολόγων που προσπαθούσαν να αποφασίσουν κάτι ε, ήταν και ο Κέινς, θα υπήρχαν ας πούμε τρεις απόψεις και άλλη μία του Κέινς. Games. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη η συμφωνία. Ελπίζουμε λοιπόν ε, η Ευρώπη να πρωτοστατήσει ε, στον αγώνα αυτό της μείωσης της φτώχειας ε, στον κόσμο και υπέρ της ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ενθουσιώδη σας τοποθέτηση. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Thank you very much for... Ευχαριστώ που μου το λόγο. Θα ξεκινήσω επενώντα αυτό το έγγραφο, γιατί για έναν επίτροπο είναι πολύ χρήσιμο να μελετά ένα τέτοιο έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις προκλήσεις και όλα τα προβλήματα και ελπίζω να μπορέσουμε με το Think Tank σας να έχουμε και πιο λεπτομέρεια ανταλλαγή απόψεων. Εγώ για μένα ανησυχώ. Στα, προηγούμενα καθή, στα προηγούμενα καθήκοντά μου ήταν και, τα προηγούμενα καθήκοντά μου περιλάμβαναν και τον Υπουργό Οικονομικών. Ε, ως Υπουργός Οικονομικών λοιπόν ε, δεν ασχολιόμουν συνήθως με αυτά τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε πάντα ως υπουργός Οικονομικών προσπαθούσα να βρω λύσεις για κάποιες ε, υποθέσεις που το άξιζαν. Και για την αναπτυξιακή πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική είναι μία από αυτές. Όλα όσα λέτε είναι σημαντικά και όντω πρέπει να πάμε και να δαπανίσουμε τα, χρώματα, τα χρήματα. Βέβαια, ο δημοσιονομικό κανονισμό δεν μου επιτρέπει και μεγάλη ευελιξία, αλλά τούτου λεχθέντος είμαι πραγματικά συμπερδεμένος για το τι ακριβώ προσπαθούμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να, όντως να έχουμε νέες, ε, νέα ξεκινήματα με αυτέ τι νέε προκλήσει. Πρέπει να ξέρουμε πού είναι ο πυρήνας της ε, υπόθεση. γιατί εδώ πέρα έχουμε επικεντρωθεί σε πολλά σημεία. Είναι σημαντικό το πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα μετρήσουμε την πρόοδο και προσπαθώ να δω εγώ τι θα ήθελα να επιτύχω. Θα ήθελα λοιπόν κάθε ένα στον κόσμο αυτό να έχει ένα άξιο βιωτικό επίπεδο. Να έχει, κάτι να, να έχει μια δουλειά, να έχει κάτι να φάει, να έχει ένα σπίτι. Αυτά είναι πράγματα που θα ήθελα εγώ να συμβαίνουν στον, στον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και μετά, προσπαθώ να σκεφτώ. Εγώ τα έχω αυτά. Ναι, θα έλεγα. Χαίρομαι που ζω στη χώρα μου. Ξέρω ότι θα έχω δουλειά. Ή τέλο πάντων κοινωνική υποστήριξη αν δεν έχω δουλειά. Και, με την ε, χώρα... και μ' αρέσει η χώρα μου παρόλο που έχει ασταθεί κυβέρνηση, έχει προβλήματα. Μ' αρέσει. Και Βασικά τι είναι αυτό που μας απασχολεί. Είναι η διακυβέρνηση. Εμπιστεύομαι τη διακυβέρνηση που γίνεται στη χώρα μου. Ότι εντάξει θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές, θα υπάρξουν και καλές στιγμές όμως, αλλά ξέρω ότι η κυβέρνηση θα νοιάζεται για τα δικά μου δικαιώματα ως μέλος της κοινωνίας. Και μετά σκέφτομαι ότι όλες οι πολιτικές που θα πρέπει να εμφωνήσουμε θα πρέπει να προέρχονται από αυτό, από το θέμα της διακυβέρνησης. Γιατί στο τέλος τέλος θέμα διακυβέρνησης είναι που πρέπει να ξεκινάει και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Γιατί από, από πάνω προς τα πάνω σημαίνει, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων και πρέπει να δικαιολογήσουμε πώς τα δαπανούμε και σε ποιους σκοπούς. Και απ' την άλλη, ποτέ δεν μπορεί κανείς να περιμένει επιτυχία σε κάποιες χώρες εάν δεν το δέχονται οι κυβερνήσεις. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να τα συνδυάσουμε αυτά και αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και είναι σημαντικό οι προσπάθειές μας να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση δεν προσπαθούμε να αποκλίνουμε από τον στόχο μας, να παρεκκλίνουμε από τον στόχο μας. Ε, γι' αυτό θα έχουμε και τα εθνικά έγγραφα στρατηγικής, τα οποία θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο στοχοθετημένα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι η ώρα που θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. για την αναπτυξιακή πολιτική λοιπόν ε, σήμερα είναι σαν να προσπαθούμε να τα καλύψουμε όλα σε όλους του τομεί. Μιλούμε για εμπορική πολιτική για, την, ε, για τις μπανάνες ας πούμε. Πάλι χρησιμοποιούμε την αναπτυξιακή πολιτική. Μιλούμε για, την, ε, για τις κλιματικές αλλαγές. Πάλι πέφτει στο τραπέζι η αναπτυξιακή πολιτική. Παντού μιλούμε για την αναπτυξιακή πολιτική. Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει, αλλά στο τέλο. Ε, πρέπει να δούμε και την αναπτυξιακή πολιτική στο δικό της πλαίσιο. Να μην τη θεωρούμε πάντα ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει τον καθένα να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Είναι και αυτή μια πολιτική από μόνη της και αυτή είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Να έχουμε δηλαδή σαφείς στόχους, σαφή πολιτική, μακροπρόθεσμη, που να έχει συγκεκριμένους στόχους, και αυτό να γίνεται με κάποια συγκεκριμένα εργαλεία. Σέβομαι όλε τι συζητήσει που έχουν γίνει για τι εξωτερικέ δράσει, για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και πώ θα, εκπροσω... πώς θα συνδυαστούν οι εργασίες που γίνονται και από πλευράς ε, γενικών διευθύνσεων και από πλευράς ε, επιτρόπων. Αλλά αυτό που προετοιμάζουμε τώρα, νομίζω ότι μάλλον ο επόμενος Επίτροπος Ανάπτυξης και η επόμενη Κομισιόν είναι αυτή που θα το ολοκληρώσει, γιατί έχουμε και χρονικούς περιορισμούς, έτσι. Και επίσης αυτό που ξέρω για την αναπτυξιακή πολιτική είναι ότι δεν είναι πολιτική για ένα χρόνο ή για έξι μήνες ή για δύο χρόνια. Είναι μια βασική πολιτική όπου θέτουμε στόχους, μετρούμε, προσαρμόζουμε, αλλά δεν αλλάζει κάθε εξάμεινο η πολιτική, ούτε οι στόχοι της και κάθε χρόνο. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό. Τούτου λεφθέντος, να έρθω στα θέματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά και για την Ευρώπη και για τα think tanks, τα οποία δεν, το έχουν, δεν έχουν σοχληθεί πάρα πολύ με αυτό. Είναι η δέσμευσή μας. Αν θέλετε μια κοινωνία που να μπορεί να επιτύχει ε, τους ε, στόχου τη, αλλά πρέπει να έχει και τα ε, οικονομικά μέσα για να το κάνει αυτό. Και υπάρχει και το θέμα του 0,7, το οποίο επίσης γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Γιατί εμείς ε, πιστεύουμε σε αυτή την πολιτική που εκπονούμε ή όχι θα μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει και στο 0,3, 0,2, 0,0 κάτι. Δεν είναι το 0,7 το θέμα. Αλλά εφόσον δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε, είναι περισσότερο ε, ηθικό πρόβλημα παρά αριθμητικό. Δηλαδή, 2 δισεκατομμύρια παραπάνω δεν θα, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Το θέμα είναι να έχουμε μια σαφή δέσμευση. Όχι απλώς, να, δεν βρήκαμε απλώ έναν άλλο τρόπο να δαπανίσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό στο αερινό πακέτο θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με ήπιο τρόπο, με ήπιο τρόπο δηλαδή πιστεύοντας την αξιοπιστία ότι η Κομισιόν δηλαδή δεν θα πρέπει να επιβάλλει τα εργαλεία αλλά αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να γίνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα κράτη-μέλη θα πούνε ότι να και άλλοι δεν το έχουν επιτύχει, η Κομισιόν θα πει να εσεί δεν τα καταφέρατε, το Κοινοβούλιο επίσης θα μας κατηγορήσει, χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, θέλουμε να συμβεί αυτό. Όχι. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά, κάτι άλλο σημαντικό. Η συνεργασία. Αποτελεσματική συνεργασία. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Το κάναμε αυτό στην ΑΕΤ. Η ΑΕΤ ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα. Γιατί εντάξει, ήταν αρκετά συγκινησιακό το όλο περιβάλλον σε ό,τι αφορά το τι έγινε στην ΑΕΤ. Όλοι δεσμευτήκαμε και είπαμε ας τα καταφέρουμε λίγο καλύτερα από ό,τι συνήθως. Οπότε, όντως, κάναμε μια, μια, μια κατανομή των ευθυνών και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον τρόπο αυτό. Γιατί αν παρεκκλίνουμε, τότε και πάλι κάνουμε καλυστία. Ποιος είναι ο καλύτερος Πάροχο αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ω παγκόσμια κοινότητα να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και για την κλιματική αλλαγή ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε ε, αν δεν μπορούμε εμείς μεταξύ μας να συμφωνήσουμε για αυτό που θέλουμε να πείσουμε τους άλλους. Για την κλιματική αλλαγή λοιπόν η Ευρώπη των 27 συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που έχουν καλό μητρό σε ό,τι αφορά τα, τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή, θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει μια απόφαση μαζί με τις χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιες ε, προκλήσεις. Η Πολωνία, ας πούμε, η Πολωνία έχει, ε, είναι μια τέτοια χώρα που μπορεί να βοηθήσει σε ό,τι αφορά την πολιτική αυτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η δέσμευση. Η Πολωνία ε, θα έπρεπε να ξέρει ποια είναι, ποιες είναι οι απαιτήσει για να αλλάξουν, οι, να αλλάξουν οι πολιτικές μας. Μετά, κάτι άλλο που είναι σημαντικό, αλλά είναι ένα καλό σημείο κίνησης. Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν μας έχουν βοηθήσει να φτάσουμε στο στόχο μας. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και οι ιδέες που υπάρχουν εδώ σε αυτό το βιβλίο και στην έκθεση του Μεσολαβητή, ε, στην αρχή ε, δεν ήμουν πολύ σίγουρος, δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες υπηρεσίες, καινούριου θεσμούς. Ο, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε, ειδικά στους τομείς που σας ανέφερα, για την ανάπτυξη δηλαδή να δούμε τι λένε και τα think tanks, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, πού πάμε για να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί από πολιτικής πλευράς όλα είναι σημαντικά, αλλά όντως πρέπει να ε, επικεντρωθούμε σε αυτό που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε καλύτερα το στόχο μας. Έχουμε προχωρήσει αρκετά και η κοινότητα ήταν αυτή που έκανε την διαφορά γιατί δεν φοβόμαστε τα στα κράτη πια. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Μάθαμε πολλά. Και τα πολλά χρήματα δεν σημαίνουν πάντα ότι βοηθούν, ας πούμε, για το Πακιστάν. Περίπου 400 εκατομμύρια πήγαν για τις δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά 10% Τη ανάπτυξη αυτή πήγε για, στην Ασία το, το Ήταν το 10% που δώσαμε στην Ασία, το 25% πάει στο Αφγανιστάν. Και προσπαθούμε να καλύψουμε α, τον κόσμο. Μήπως όμως πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες συγκεκριμένε χώρες. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κενά στην, στην πολιτική μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Και ένα τελευταίο για την κατανομή των ευθυνών σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Είναι ατυχής γιατί ε, μόνο τον προγραμματισμό σκέφτεται και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Ο προγραμματισμός πάντα μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά αν είναι αυτό το μόνο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, μάλλον κάτι δεν πάει καλά σε αυτό που συζητάμε. Βεβαίως αργότερα αν θέλετε μπορώ να πω και κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο φλεγόμενο θέμα και θα έπρεπε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μια μεγάλη ισχυρή υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, όχι όμως εις βάρος της ενδεξιακής πολιτικής, αλλά για να την ενισχύσει. Το λόγο τώρα έχουν οι κυρίες ευρωβουλευτές. Κυρία Ντέβα, καταρχήν. Πρόεδρε. Στις 5.30 ε, σήμερα το απόγευμα πραγματικά ενθουσιάστηκα. Ε, είχαμε εδώ τέσσερις προσώπους των δεξαμενών σκέψεων που μας παρουσίασαν νέες ιδέες για την ανάπτυξη, για τη μείωση της στόχης ε, σε όλο τον τομέα στον οποίο εργαζόμαστε. Και τι άκουσα τελικά άκουσα το ίδιο πάντρα, το ίδιο δόγμα. Δηλαδή, τι το καινούργιο υπόθηκε τώρα. Μπορούμε ένα λεπτό να σταματήσουμε και να σκεφτούμε και να αναρωτηθούμε αν οι ακόλουθες χώρες έγιναν πλούσιες λόγω των πολιτικών που ακούσαμε. Έχουμε ακούσει την ε, πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα της βοήθεια, ανάπτυξη χαμηλού άνθρακα, ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ε, αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Σουηδία και η Φιλανδία, παραδείγματο χάρη. Έγιναν πλούσιες χώρες λόγω όλων αυτών που ανέφερα. Και σκόπιμα χρησιμοποιώ αυτές τις χώρες, γιατί θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες χώρες ε, ε, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιε τέτοιες χώρε όπω ε, η χώρα που γεννήθηκα. Όμω μήπω εδώ κάτι δεν καταλαβαίνω, γιατί από ό,τι φαίνεται να είναι σε μένα προφανέ. δεν είναι προφανέ. Στου Ευρωπαίου εγώ έρχομαι από μια φτωχή χώρα σε μια πλούσια χώρα και να ρωτιέμαι πώς έγιναν πλούσιοι οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έγιναν πλούσιοι κάνοντα κάτι από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έγιναν πλούσιοι λόγω τη δημιουργία του πλούτου wealth creation και πουθενά σε αυτή την έκθεση δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Δεν μπορεί κανείς να εξελίψει τη φτώχεια χωρίς να δημιουργήσει εργασία. Χωρίς να δημιουργήσει πλούτο. Η Κίνα σημείωσε μάλλον τρία 300 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια και 200 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είναι πλέον φτωχοί γιατί δημιούργησαν πλούτο και βγήκαν από την παγίδα της φτώχειας. Και υπάρχουν 9-3 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων εκεί έξω σε αναπτυσσόμενες χώρες που δεν αποτελούν τμήμα των νόμιμων οικονομιών των χωρών αυτών. Όμως ποτέ δεν βγαίνει εδώ, ποτέ δεν εξτομίζουμε εδώ τη φράση δημιουργία πλούτου δεν λειτουργεί όλο αυτό. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες καινούριε ιδέες. Κυρία Κέλλερ παρακαλώ. Νομίζω ότι θα προχωρούσαμε κάπως παραπέρα αν εφαρμόζαμε ήδη όσα αναφέρατε στην εκθεσή σα, δηλαδή τη συνοχή της πολιτικής. Έχουμε πάρα πολλές αντίθετα και θέλουμε να υπάρξει υπέρ όλων αυτών, αλλά αν δείτε τι γίνεται στην πράξη, βλέπουμε τα αντίθετα και θέλουμε να υπάρξει αλλαγή τη πολιτικη όχι περαιτέρω δηλωσει και διακηρύξει. Αν δούμε λόγω χάρη την ελευτική πολιτική, την αγροτική πολιτική, ξέρουμε ακριβω που είναι τα προβλήματα, αλλά δεν τα αλλάζουμε. Θα ήθελα πάντως ε, να σας συγχαρώ για αυτή την πολύ καλή έκθεση και σας ευχαριστώ γιατί συμφωνήσατε με πολλά με το όσο είπα εγώ στη δική μου έκθεση για την ε, πολιτική συνοχής. Υπάρχουν κάποια θέματα που αναφέρετε στην παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε στο ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχει το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Αν, παραδείγματο χάρη, σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε τη διμερή, τα διμερή συστήματα ε, για την ε, χορήγηση βοήθεια, τα ε, χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, δεν ήταν καλύτερο να έχουμε χορήγηση βοήθεια μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης Αναφερθήκατε στο προγράμματα, ε, αλλά τι θεωρείτε ότι είναι ζωτικό, ποια θεωρείτε ότι είναι ζωτικά καθήκοντα του Επιτρόπου Ανάπτυξης και τι θεωρείτε ότι πρέπει να περάσει στην κυρία Άστον. Θα ήθελα την άποψή σας από αυτό. Επίσης, ε, κάνατε κάποιες προτάσεις για μηχανισμούς ε, συνοχής πολιτικών στο εσωτερικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, πώς ε, θα μπορούσε να γίνει η παρακολούθηση και χάρηκα επίσης που υποστηρίξατε την ιδέα του διαμεσολαβητή ως μια δυνατότητα προσφυγής, κατάθεσης προσφύγων, όμως επειδή μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με την ιδέα αυτή, εσείς μπορείτε να μας πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι το πλεονέκτημα να έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό κατάθεσης προσφυγών ή παραπώνων, αν θέλετε, στον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκέρεντ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που έλειπα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, οπότε θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτά που άκουσα Θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες ε, παρεμβάσεις του Επιτρόπου σε σχέση βέβαια με αυτά που άκουσε. Η συνένεση, το έγγραφο συνένεση για την ανάπτυξη υπάρχει, έχει μία φράση που λέει ότι είναι αυτοσκοπός η αναπτυξιακή ε, συνεργασία και είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο σε όλους όσους δούλεψαν για την έκθεση αυτή. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε Γι' αυτό το βασικό θέμα, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε τη συζήτηση. Όλοι όσοι έχουν αρμοδιότητα για την αναπτυξιακή συνεργασία θα έπρεπε να μας πούνε ποια είναι η άποψή τους για το θέμα αυτό, ποια είναι, ποιο είναι το στρατηγικό τους όραμα, ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους όταν ζητούν αρμοδιότητες. Δεν έχει νόημα να συζητάμε έτσι γενικώς και αορίστως για τις αρμοδιότητες, πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές. Θα ήθελα λοιπόν όλες τις απόψεις εγώ να τις ακούσω. Διαφορετικά δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να γυρίσουμε στα βασικά. Και δεν μπορώ να πω και περισσότερα γιατί ένα μεγάλο τμήμα της συζήτηση. έλειπε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Äh, ναι, πρόεδρε. Θα πω απλώ ότι όντω είναι δύσκολο να κάνουμε έτσι μια σύνοψη των απόψεων όλων των εμπλεκομένων και να συμφωνήσουμε επί κειμένου. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι έχω την αίσθηση ότι κάποια ερωτήματα δεν συζητηθήκαν πολύ. Λίγο συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης του πληθυσμού, της αύξησης του πληθυσμού. Ε, είναι πραγματικά δραματικό θέμα σε ό,τι αφορά τη δουλειά που θα κάνουμε και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Επίσης, πάρα πολύ λίγο. Επίσης, πάρα πολύ λίγο έχουμε συζητήσει τι είναι εφικτό από όλους αυτούς τους στόχους της χιλιετίας που έχουμε θέσει και τι θα ήταν ευκταίο Νομίζω αυτόν τον ε, ισολογισμό θα μπορούσαμε να τον ε, κάνουμε για να μπορέσουμε έτσι να επιτύχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη ε, και επίτευξη τελικά των στόχων μας. Επίσης, ένα θέμα που συζητείτε συχνά στο θέμα της αναπτυξιακής πολιτικής είναι το ότι ζητάτε, ζητούνται συνέχεια περισσότερα χρήματα. Κατανοητό αυτό, γιατί είναι και η εύκολη λύση. Αλλά νομίζω ότι ελάχιστα έχουμε συζητήσει. Γιατί, για παράδειγμα, σε πολλές ασιατικές χώρες πέτυχαν να βοηθηθούν από, τη, από τις δικές τους δυνάμεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία απάντηση σε αυτό. Και επίσης, ελάχιστα έχει συζητηθεί το θέμα της επικουρικότητας. Εγώ όταν μιλώ με, με εμπειρογνώμονες από τη δική μου την χώρα, από τη Γερμανία, εμπειρογνώμονες περί τέτοιων θεμάτων, υπάρχει μεγάλη κριτική έναντι των μέτρων που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι από ανθρώπους που είναι φορείς και εμπλέκονται, αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν επιτόπου την κατάσταση και ξέρουν πού πάνε τελικά αυτά τα κονδύλια. Τέλος, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του καλύτερου συντονισμού Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα καυτά ερωτήματα και θα ήθελα περισσότερες και πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να θέσουμε και σε εσά ερωτήματα, κύριε Επίτροπε. Ίσως να μην το άκουσα. Μπορείτε να μας πείτε εσείς κάτι για την οργάνωση της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων, για τις λειτουργίες της, για του τομεί για, την οποία, για τους οποίους, στους οποίους εμπίπτει και η αναπτυξιακή βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που είναι, παρίσ... που είναι παρόν ε, στην ε, σημερινή μας συνεδρίαση. Εχθές είχε, είχε έρθει η κυρία Γεωργίευα συζητήσαμε μαζί της ε, τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με ανθρωπιστική βοήθεια και ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να το πω γιατί ελπίζω το ίδιο να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει και για το οποίο μιλήσατε κάπως και την προηγούμενη φορά το είχατε αναφέρει για τα υπερπόντια διαμερίσματα. Υπήρξε μια ανακοίνωση τον Νοέμβριο και παρουσιάστηκε μια στρατηγική για τις άκρος απομονωμένες περιοχές, δηλαδή μια δουλειά για την ανταγωνιστικότητά τους και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Θα ήθελα να μας πείτε ποια θα είναι η στρατηγική σας σε σχέση με τα με τα υπερπόντια διαμερίσματα. Έχετε σκοπό, και μιλάω για τη Νέα Καλλιδονία για παράδειγμα, μήπως θα μπορούσατε να θεωρήσετε για παράδειγμα ότι θα μπορούσε να είναι μία βασική περιοχή από την οποία θα ξεκινούσαν οι δραστηριότητε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα. Μήπως θα μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιηθούν κάπως σαν προπύργια ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό εντάσσεται στην δική σας στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Λεβίν, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική στο να αλλάξουμε και να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε όλους τους τομείς προκειμένου να συνάδουν με τις αναπτυξιακές πολιτικές. Αν δούμε λόγου χάρη τι συμβαίνει στην Αλία, στη Γεωργία ή στο εμπόριο, στις σχετικές πολιτικές, είναι προφανές ότι αν επιτρέπουμε στις ευρωπαϊκές ε, τράτες ε, να αλλιεύουν όλα τα ψάρια στη Δυτική Αφρική, τότε ε, τελικά θα πρέπει φυσικά να προσφέρουμε κάποιε θέσει εργασία στου Ελλήνε που δεν μπορούν να ψαρέψουν τα δικά του ψάρια. Αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα παραγωγικό. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει καταρχήν ε, να εξετάσουμε τις δικές μας πολιτικές προς πάσα κατεύθυνση. Μα... πάρα πολύ η δήλωση του Επιτροπού Πίμπαλξ Θεωρώ ότι ήταν ένα ε, καλό τρόπος να παρουσιάσετε τι πραγματικά χρειάζεται και καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι είναι βασική διακυβέρνηση και ότι κάθε προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται προ αυτή την κατεύθυνση. Μόλι ε, επέστρεψα από μια αποστολή παρατήρησης εκλογική διαδικασία στο τοκό. Το και προσπάθησα να καταλάβω όλα τα τεχνικά στοιχεία και όλες τις ε, θεσμικές δυσκολίες ε, ε, που ενέχονται στην υλοποίηση δίκαιων εκλογών. Υπάρχουν δυσκολίες και επειδή πολλοί άνθρωποι είναι ανελφαβήτοι και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις πολιτικές συζητήσεις και έχουμε στρέβλωση από τα ΜΜΕ όπου ο πρόεδρος κατέχει το 95% του χρόνου στα ΜΜΕ. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν ο νέος Επίτροπος έχει κάποιες ιδέες για το πώς ε, θα ε, προσφέρει προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ο νέος Επίτροπος κάποια ιδέα σε σχέση με το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι η διακυβέρνηση είναι πραγματικά βασικό θέμα, γιατί αν δεν έχουμε θεσμούς που να λειτουργούν καλά στις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, τότε δυστυχώς ε, η βοήθεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει. Κύριο Χάρλεμ ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, ε, κύριε Επίτροπε, η εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη χρηστή διακυβέρνηση της χώρας μας είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών και το πραγματικό κοινό καλό και κοινό αγαθό που έχει ο κάθε ε, άνθρωπος είναι η πολιτεία, το κράτος του οποίου η διαχείριση είναι διαφανής. Όταν βλέπουμε την κρίση στην ΑΕΤ, για παράδειγμα, μετά από το σεισμό και το συγκρίνουμε με το τι έγινε στο στη Χιλή, η ίδια δραματική κατάσταση δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα στη μία χώρα και στην άλλη. Και θα μπορούσαμε αυτή, αυτόν τον προβληματισμό να τον επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των think tanks αν πιστεύουν ε, ότι η αναπτυξιακή συνεργασία έχει βοηθήσει την οικοδόμηση των κρατών που είναι η βάση μιας ε, πολιτικής ανάπτυξης ε. αυτοί που πέτυχαν, είπε ο κύριος Ντέβα, ήταν εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν πλούτο. Υπάρχει όμω και μία άλλη πτύχη και αυτό έχει να κάνει με τη σχέση τη εμπορική και τη αναπτυξιακή πολιτική μα. Ε, μία προσπάθεια όχι μόνο καλή τοποθέτηση οικονομική ε, στο πλαίσιο τη ε, κατανομής εργασία, αλλά και οικονομική διαφοροποίηση, ώστε να μην υπάρχει έκθεση στην υπερπαραγωγή, για παράδειγμα. Και γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να μου απαντήσουν και τα think tanks, να μα πούνε λίγο περισσότερε λεπτομέρειε σε σχέση με το εμπόριο δηλαδή εμπορικέ πολιτικές μας ε, στις χώρες ε, ΑΚΕ ή σε άλλες χώρες ε, πράγματι συνεισφέρουν στην οικονομική διαφοροποίηση που κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις βασικές πτυχές της ανάπτυξης. Ναι, γεωργία, αλλά όχι μόνο στραμμένη προς τις εξαγωγές και άλλες παράλληλες δραστηριότητες, άλλες υπηρεσίες επίσης. Να μην πιέζουμε μόνο τις χώρες εκείνες του Νότου που ήταν πρώην απικίες ε, να, τους, ε, να τις πιέσουμε σε μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή γιατί αυτά μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα. Αντιθέτως να μπορέσουμε κάπως να τους εκβιομηχανίσουμε κατά κάποιο τρόπο όπως έγινε στην Ασία. Παράλληλα όμως να υπάρχει και κάποια ε, συνειδητοποίηση της ευαισθησίας τους. Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των Think Tanks για τις ε, αναπτυξιακές μας πολιτικές του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής ε, που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο κ. Φίσας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να επιμείνω, σωστά ανέφερε η συνάδελφος Ιζαβέλα και εγώ ήμουν στο Τόγκο, στην ε, αποστολή παρατήρηση των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε αυτό το είδος των αποστολών γιατί αφενός είχαμε πολλές επαφές ε, με τον πληθυσμό και αισθανθήκαμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη ε, στήριξης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολλοί νέοι μας έλεγαν ότι έχουμε κουραστεί από την ξύλινη γλώσσα, και πραγματικά αυτό ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη για τους ανθρώπους που ζουν εκεί και εξοδεύουν τόσα χρήματα. Αλλά από την άλλη, ε, ίσως ε, θα μπορούσε και η αντιπολίτευση να χρησιμοποιήσει κάποια μέσα ε, για να οργανώσει διαδηλώσεις που μπορεί να είχαν πολύ σημαντικές ε, Συνέπειε, Δηλαδή εδώ βρισκόμαστε μεταξύ δύο πυρών. Τι να κάνουμε, να πούμε την αλήθεια για τα πάντα ή να μην την πούμε για να αποφύγουμε ε, τα χειρότερα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώ οργανώνονται αυτές οι αποστολέ. και σε ορισμένε περιπτώσεις ε, θα πρέπει να βλέπουμε αν πληρούνται οι ελάχιστες εγγύσεις για να μπορέσουμε να τις υλοποιούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εαυτό μου και να πω ότι το θέμα της διακυβέρνησης ε, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ και έχω εργαστεί πάρα πολύ στο ζήτημα αυτό. Και πολλές φορές έχουμε απέναντί μας ε, την αρχή της ε, κυριαρχίας των κρατών. βλέπουμε ότι πολλές φορές οι ηγέτες ορισμένων χωρών τις λαιλατούν και πραγματικά είναι ιδιαίτερη επιτυχή στο να κρύβουν ε, τη ηλία τους, τα λάφυρά τους και πολλές φορές χρησιμοποιούν και τις δικές μας τράπεζες και τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ε, κακή διακυβέρνηση αν συνεχίζουμε να ανεχόμαστε την ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων και των μυστικών δομών που επιτρέπουν και στις πολυθυμικές να μην πληρώνουν φόρους και στους διαφραγμένους ηγέτες να ε, έχουν διευκόλυνση να λαιλατούν. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώπιον ε, αυτού του φαινομένου είμαστε αρκετά αδύναμοι, προσπαθούμε να το παρακάμψουμε. Εγώ προσωπικά προσπάθησα να συνδράμω ε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε αρκετές χώρες, χρηματοδοτήσαμε εμπειρογνωμοσύνη για να δούμε τελικά τι, ότι όταν γίνονταν λειτουργικές ε, ε οι λειτουργικοί αυτοί οι οργανισμοί τότε οι οργανισμοί αυτοί ήδη ε, όταν αποτελούσαν απειλή, τότε τους διέλυαν. Αυτό ε, έγινε στην Ιγυρία, έγινε στην Τανζανία, στη Ζάμπια. Τα αρμόδια άτομα ε, τελικά για τη διάλυση των υπηρεσιών πήραν την εξουσία τελικά και θα ήθελα να ρωτήσω ε, τους ε, συμμετέχοντες στα Think Tank αν μπορούν να ξεύρουν μία λύση σε αυτό το θέμα. Και το λόγο έχει τώρα ο κύριος ε, Πίμπαλξ για να κάνει κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Πρόεδρε, έχω λίγο μπερδευτεί γιατί τα Think Tanks νομίζω ότι θα πρέπει να πούνε τη δική τους άποψη. Γιατί εγώ έχω έρθει, θα ξανάρθω στην Επιτροπή σας. Δεν θέλετε να μιλήσετε πρώτος. Ε, να πω ένα πράγμα που είναι σημαντικό. Μάλλον δύο πράγματα. Καταρχήν σε σχέση με την ε, υπηρεσία της Κομισιόν για τις εξωτερικές, για τις εξωτερικές δράσεις. Μέχρι στιγμή ακόμη δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, οπότε είναι δύσκολο να σα απαντήσω σε αυτό που θέλετε για την υπηρεσία αυτή. Αλλά ούτω ή άλλω, ό,τι προταθεί θα πρέπει να βασιστεί στο γράμμα και το νόμο της, ε, στο γράμμα και το πνεύμα της συνθήκης της Αβώνας Πρέπει να έχουμε μία ενιαία φωνή όταν παρουσιάζουμε τους στόχους μας και τις δράσεις μας στην εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι σαφές και το συμμερίζομαι απόλυτα. Η συνθήκη λέει ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι πολιτική από μόνη της. Δεν είναι πολιτική ε, ε, ε, συμπληρωματική στις εξωτερικές δράσεις που καμιά φορά τη χρησιμοποιούμε και καμιά φορά όχι, η αντιμετώπιση τη φτώχεια είναι ας πούμε ένα συγκεκριμένο στόχο αυτή τη πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα εκπονήσει τον προπολογισμό της η Κομισιόν. Και επίση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ω βάση και την παρελθούσα εμπειρία ώστε να υπάρξουν σχέσει μεταξύ των δραστηριοτήτων τη υπηρεσία και των δυναμικών που έχει η Κομισιόν. Οπότε δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή. Μπορεί να γίνει με διάφορου τρόπου αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι οι αρχέ που θα πρέπει να καθοδηγήσουν την τελική μα απόφαση. Και για να κλείσω. ποιε είναι οι δικέ μου, απαιτήσει, από, του, από τα think tanks. Προσπαθούν έτσι να μας πιέσουν, γιατί στην αναπτυξιακή πολιτική νομίζω ότι πολλές φορές τα νερά είναι ήρεμα. Και ήδη υπάρχουν πολλές προσπάθειες που γίνονται. Σημαντικό είναι να υπάρξουν αυτές οι πρωτοβουλίες και μέσω του Κοινοβουλίου και είναι καλό να συζητάμε γιατί, εντάξει, δεν συμφωνούμε όλοι, δεν έχουμε όλη την άποψη. μπορεί να μην συμφωνείτε μαζί μου, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και το σημαντικό είναι να συνεχίζεται ο διάλογος. Και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε όλα όσα γίνονται μέχρι στιγμή και ταυτόχρονα να τα βελτιώσουμε. I now give the floor to Mr. Maxwell. Ο κύριος Μάξουελ έχει το λόγο για να συνοψίσει εκ μέρους των Think Tanks. Στις 5.39 νόμιζα ότι δεν πάει πολύ άσχημα το πράγμα. Και μετά μας είπανε ότι τίποτα δεν έχουμε κάνει, ότι τα πράγματα έχουν παραμείνει ίδια. Κάποια όντω έχουν παραμείνει, αλλά ειδικότερα για το θέμα το οποίο θέσατε, συμφωνούμε με την ανάπτυξη, συμφωνούμε με τον ιδιωτικό τομέα, με αυτό που είπατε για τον ιδιωτικό τομέα, και είναι από τα βασικά μα κεφάλαια, που δεν αναφέρεται όμω το Ευρωπαϊκό Έγγραφο για την, τη συνένεση για την αναπτυξιακή βοήθεια. Κοιτάξτε, ποια είναι η ευρύτερη εικόνα. Νομίζω ότι του χειρότερου ε, κινδύνου αποφύγαμε. Ο μεγαλύτερο μου φόβο ήταν, ε, θα ήταν, ότι, ήταν ότι ο Επίτροπο Πίμπαλξ δεν ε, θα μπορούσε να έχει ε, να μπορεί να ελέγξει την ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια και το λέω αυτό ως άνθρωπος που 12 χρόνια συμμετέχει σε ένα think tank και πάντα πίστευα ότι δεν θα είμαι ποτέ κάτι παραπάνω από διευθυντής ενός think tank και χαίρομαι που εσείς κύριε Επιτροπέ δεν είστε σε αυτή τη θέση γιατί έχετε τη γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και τη EuroPaid ε, και μπορείτε τουλάχιστον να βασιστείτε στην ε, εφαρμογή των βασικών μέσων. Αλλά όταν πηγαίνεις ας πούμε σε σεμινάρια κάποιο σου λέει ποια, ποιες είναι οι ανησυχίες σου για το μέλλον. Εγώ πέντε τουλάχιστον ανησυχίες έχω και σε κάποιο βαθμό ε, νομίζω ότι θα εξακολουθήσω να την έχω. Νομίζω ότι έχουμε γραφειοκρατία χωρίς αξίες, μετά ότι θα έχουμε χρήματα χωρίς πολιτική θα επικεντρωνόμαστε στα εθνικά και όχι στα παγκόσμια. Θα είχαμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς τα κράτη-μέλη και ο πέμπτος φόβος, και δεν είναι καινούριο αυτό, ότι θα είχαμε λόγια χωρίς πράξεις. Αν λοιπόν πάρει κανείς τους φόβους αυτούς ε, και προσπαθήσει να τους κάνει φιλοδοξίες, έχει πολλή δουλειά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και ο γνώμονας πρέπει να είναι οι αξίες ε, της παγκόσμιας κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όλοι όσοι τα αναφέρατε μας βρίσκεται απολύτως σύμφωνος. Τώρα όσον αφορά τα ζητήματα, όχι, και πολιτική δέσμευση χρειαζόμαστε, όχι μόνο χρήματα. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι μίλησαν ε, για ευάλωτα κράτη, για ε, διαφθορά. Μιλάμε για μια ικανότητα πολιτικής ανάλυσης και μια ικανότητα πολιτικής παρέμβασης όταν ε, υπάρχει ανάγκη. Ναι στο εθνικό, αλλά ναι και στο παγκόσμιο. Όλο λέμε ναι πρέπει η εκπαίδευση, πρέπει οι συστήματα υγείας ε, για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, αλλά μετά δεν υπάρχει κανένα συντονισμός ε, και όλα καταραίουν. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή ηγεσία και για τα κλιματικά ζητήματα και στο G8 και στο G20 και σε, πολλά άλλα, ε, σε πολλές άλλες σημαντικές συναντήσεις μέχρι το 2012. Ευρώπη, και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα μέσω της Ευρώπης, ναι βεβαίως και θα έπρεπε. Γιατί μόνο 20% των δαπανών μας περνούν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μειώνεται ο αριθμός αυτός, γιατί έχετε παγιδευτεί με μέσα τα οποία δεν σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε το γεγονός ότι αυξάνεται η βοήθεια. Και τέλος, και αυτό βέβαια αφορά τα επιτόπου αποτελέσματα και δεν μιλάω εκ μέρους άλλων, για τη δική μου χώρα μιλάω, είναι πολύ δύσκολο να πουλήσει κανεί την, την ανάπτυξη όταν ε, έχει, υπάρχουν ε, περικοπέ στι δημόσιε δαπάνε και ε, φορολογικέ αυξήσει. γιατί είναι σαν να παίρνουμε λεφτά από τους σχετικά φτωχούς για να, τους δώσουμε σε, να τα δώσουμε σε ανθρώπους που είναι ακόμη φτωχότεροι σε άλλες χώρες. Είναι δύσκολο να το πουλήσουμε αυτό και πρέπει να μπορούμε να δείξουμε αποτελέσματα να το κάνουμε. Ναι, έχουμε πάθος για την Ευρώπη, αλλά είμαστε και εξαγριωμένοι γιατί ε, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που τα λατρεύω, αλλά 55% των χρημάτων πηγαίνουν σε μη φτωχέ ε, Αυτό είναι διάκριση κατά των φτωχών και δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της διαφθοράς ε, και για τα θέματα της λαιλασίας για τα οποία μιλήσατε, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που δεν λειτουργούν σε σχέση με τις διάφορες, με, για τη σχέση μεταξύ των γενικών διευθύνσεων ενδεχομένως. Έχουμε ένα πρόβλημα να λύσουμε και τώρα πρέπει να το λύσουμε. Είναι η στιγμή να το λύσουμε. Είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε να είμαστε κάπως πιο... Ε, να, να, να παρουσιάσουμε μεγαλύτερε προκλήσεις κύριε Επίτροπε την επόμενη φορά και όταν δεν συμφωνούμε με διάφορα πράγματα θα σας το λέμε κάθε φορά. Πραγματικά έχετε να σκαρφαλώσετε πολύ μεγάλο βουνό, αλλά όταν θα φτάσετε θα σας ανταμείψει. Έχουμε 25 ακόμη λεπτά, λέει η Πρόεδρος. Καταπληκτικό. Οπότε μπορείτε να πάρετε το λόγο. Η κυρία Κέλλερ και ο κύριος Ντέβα θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε ας ξανασυζητήσουμε. Thank you. Um, Ashley, my question wasn't uh, whether we should put more Το ερώτημά μου ήταν αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό πρέπει να έχουμε περισσότερη προσοχή αλλά μόνο όχι διμερής, ε, διμερής συνεργασία για τα θέματα της ανάπτυξης με τις αναπτυσσόμενες χώρες, μόνο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Συμφωνείτε με αυτό. Και το ερώτημα του διαμεσολαβητή για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η άποψή σας. Ποια είναι η άποψή σας για τη θέση του διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια τώρα που ανταλλάσσουμε έτσι από, απόψεις και είμαστε έτσι λίγο πιο άνετα. Αν μπορώ, θα ήθελα με τους συνομιλητές μας να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πλούτο και να απαλείψουμε τη φτώχεια. Σε όλα μας τα ταξίδια στις ανατουσόμενες χώρες έχουμε δει χιλιάδες εργαστήρια όπου κάποιοι επισκευάζουν ε, ε μοτοσυκλέτες, φτιάχνουν τσάντες, ε, φτιάχνουν ζωλήνες, οτιδήποτε τέλο πάντων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα έχουμε δει στα πεζοδρόμια, στις άκρες του δρόμου, όπως πάμε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας. Πολύ, έτσι, είναι πολύ δραστήριοι και πολλή δουλειά γίνεται. Αλλά κανένας από αυτούς, καμία από αυτή τις οικονομικές δραστηριότητες δεν είναι κομμάτι του νόμιμου συστήματος είναι παράνομες όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες. Ούτε στο ΑΕΠ λαμβάνονται υπόψη, ούτε στους... Ε, δεν υπάρχει καμία καταγραφή αυτών των εταιριών, δεν μπορούν να πουλήσουν τίποτα από αυτά που φτιάχνουν σε κανέναν άλλον, εκτός από το γειτονά τους. Γιατί αν προσπαθήσω εγώ να αγοράσω κάτι, δεν θα είχαν τίποτα να μου πουλήσουν. Δεν έχουν καμία καταχώρηση, δεν έχουν βιβλία, δεν κρατάνε ούτε διπλά βιβλία δεν έχουν καμία νοοτροπία επιχείρησης όπως την ξέρουμε εμείς και δεν έχουν και καμία δυνατότητα να πάνε να δανειστούν χρήματα, να δώσουν δάνεια, να κάνουν οτιδήποτε τέλο πάντων. Αλλά αν προσθέσετε τον όγκο αυτών των επιχειρήσεων ή την αξία τους και να πείτε ότι δεν αξίζουν πάνω από 1000 ευρώ δολάρια η κάθε μια. Το σύνολο, το έχουμε υπολογίσει, και στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες και στη ΣΥΠΑ είναι 4-3 εκατομμύρια δολάρια. Παραπάνω δηλαδή από την κεφαλαιοποίηση του ε, χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Τίποτα δεν έχει γίνει όμως ώστε να γίνουν επίσημες αυτές οι παράνομες δραστηριότητε. Το ίδιο ισχύει και στις, ε, και στην ιδιοκτησία. Ξέρουμε ότι πολλοί ζουν σε παραγκουπόλεις. Κανένας πρόεδρος, κανένας πρωθυπουργό, καμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάει με μπουλντόζες και να τα ρίξει τα, ε, τις παραγκουπόλεις αυτές. Και επίσης ξέρουμε ότι αυτές οι παραγκουπόλεις θα συνεχίσουν, θα επεκτείνονται και τα επόμενα 50-100 χρόνια. Κανένα δεν έχει τίτλο ιδιοκτησία όμω κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορούν να τη βάλουν υποθήκη, δεν μπορούν να έχουν κεφάλαια πάνω στην, να κερδίσουν κεφάλαια από την ιδιοκτησία που έχουν. Αν δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τους τίτλους των ε, σπιτιών τους, έγινε στο άτσι αυτό. Ε, κατά τύχη. Φωτογράφησε η Κομισιόν τα σπίτια που τα πήρε το τσουνάμι. οι φωτογραφίες αυτές έγιναν έτσι μια, ένα, ένας τίτλος ιδιοκτησίας. Και σε κάποιους δόθηκαν αυτές οι φωτογραφίε φωτογραφίες και τους είπαν ορίστε αυτό είναι το σπίτι σας και αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να πάει να δανειστεί και να φτιάξει το εργαστήρι του που επισκευάζει μηχα, ε, μηχανές, μοτοσυκλέτες. 7 εκατομμύρια ευρώ κάθονται και δεν υπάρχει κανένας τίτλος για να διεκδικηθούν αυτά τα λεφτά. Αν μπορέσουμε λοιπόν να, να δώσουμε επίσημους τίτλους και για τις, για τις επιχειρήσεις τους και για τα σπίτια τους, θα μπορούσαν ίσως τόσα λεφτά που έχουν να έρθουν να αγοράσουν τις δικές μας τις χώρες. Το τι πώς θα γίνει αυτό είναι δική μας δουλειά you wanted the Κύριε Πίμπαλξ, ε, θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, ακούσαμε τις προτάσεις των Θεμητανικά, αλλά είχαμε και μία σαφή ερώτηση του Πόγκα γιατί ε, ρώτησε για τα υπερπόντια διαμερίσματα και δάφη. Τα πρώτα καλά νέα ναι, για μένα είναι ότι κανένα δεν μπορεί, να προσπαθεί να ε, τα αφαιρέσει από την Κομισιόν, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε μαζί τους και εγώ πιστεύω πολύ σε αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω κυρίως σε αυτόν τον τομέα. Έτσι λοιπόν θα σας πω ότι θα απαντήσω ε, σε αυτά τα απερχόντια μερισμένα. Όμως τώρα για τις νήσους του Ειρηνικού έχω μια εμπειρία με την νήσους του Σολομόντα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ουσιαστικά δύο-τρία στοιχεία ε, σε όλες τις πολιτικές μας καταρχήν είναι μικρά αλλά έχουν τα ίδια βασικά προβλήματα που έχουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να γίνει στο ίδιο επίπεδο όπως γίνεται και με τις μεγαλύτερες χώρες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και επίσης ε, δεν θα πρέπει ε, ε, θα πρέπει μάλλον να υποστηρίζουμε τη διακυβέρνηση μέσω του περιπολογισμού να λαμβάνουμε αντίστοιχα μέτρα προκειμένου να τους κάνουμε να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνοι και ταυτόχρονα να μετράμε και το output, τα αποτελέσματα, αλλά να μην δημιουργούμε υπερβολική γραφειοκρατία στο input. Και επίσης έχουμε και την ιδιαίτερη εστίαση στην κλιματική αλλαγή, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να καταβαλούμε προσπάθειες για, για το μετριασμό ε, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για τις νήσους αυτές, γιατί εκεί θα πρέπει να δοθούν τα πρώτα κονδύλια. Αυτό είναι προφανές, αυτό ήθελα να αναφέρω για να απαντήσω την ερώτηση του κ. Πόγκα. Κύριε Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω ε, και ο κύριο Γκέρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στην αρχή τη παρουσίασή σα, Βέβαια, σκοπεύω να διαβάσω εκτενώς το κείμενό σας ήδη άρχισα να το διαβάζω και φυσικά την Παρασκευή έχω και συνάντηση με τους εκπροσώπους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στο Λονδίνο. Σίγουρα θα συζητηθεί το έγγραφο αυτό. Μου άρεσε η προσέγγιση του κυρίου Μάτζουελ και θα ήθελα να πω ότι σπάνια έρχονται think tank που να κάνουν τόσο παθιασμένες παρουσιάσεις, συγχαρητήρια Επίσης, ε, να σας πω ότι εμείς ε, δεν έχουμε πρόβλημα να αναγνωρίσουν οι φτωχοί τα ωφέλη του να δίνουμε στους άλλους. Ε, η προβληματική είναι κυρίως όσοι βρίσκονται στο μεσαία και στα υψηλότερα στρώματα και το επιχείρημα στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματικά υποστηρίχθηκε στην κοινή γνώμη. Έτσι λοιπόν αυτό με οδηγεί στην ανάπτυξη και στο πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι η οριζόντια προσέγγιση είναι η μόνη προσέγγιση. Μιλάμε για συνοχή των πολιτικών. Νομίζω ότι θα πρέπει να το στρέψουμε αυτό και να πούμε ας μην έχουμε συγκρούσεις μεταξύ των πολιτικών και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν έχουμε οριζόντιες προσεγγίσεις στο να δημιουργούμε αποτελεσματική ανάπτυξη, ας ε, βγάλουμε από την εξίσωση την ε, αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ε, μιλήσουμε για όλες ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καμία χώρα δεν έχει φτάσει στην επιτεύξη του δυναμικού της, έτσι. λοιπόν, είναι ιδέα πίσω από την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, μπαίνω τώρα σε ένα καυγά κατά κάποιο τρόπο. Η ιδέα πίσω από την ανάπτυξη είναι ότι όλοι έχουμε κάτι να κερδίσουμε από αυτό, γιατί έχετε απολύτω δίκιο. Αν κάποιο έχει μία δουλειά, και νομίζω ότι ε, δεν χρειάζεται να σα πείσω για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία. Αν κάποιο έχει λοιπόν ε, μία δουλειά, αν είναι νόμιμα απασχολούμενο, καταβάλει εισφορέ και καταβάλει και φόρου, αλλά χρειαζόμαστε στη συνέχεια ορθιδία κυβέρνηση για να συλλέγονται οι φόροι και να διανέμονται Στη συνέχεια πρέπει να δούμε το θέμα των υποδομών. Πρέπει να υπάρχουν υποδομέ, γιατί μόνο η ύπαρξη θέσεων εργασία δεν λύνουν τα προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει του τίτλου τη γη, αλλά έχουμε αποχετεύσει, έχουμε πρόσβαση στα φάρμακα, στο πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει λοιπόν μια απλή απάντηση, αλλά νομίζω ότι αυτή η δέσμευση να πούμε ότι κάτι δουλεύει σε άλλε χώρε, γιατί δεν δουλεύει εδώ, μπορούμε να το δούμε αυτό. Αυτό ελπίζουμε να μα οδηγήσει προ. Ε, την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας το 2015. Και ας θυμόμαστε, δεν είναι το τέλος το 2015, είναι η αρχή. Νομίζω ότι έχουμε λοιπόν ε, μια ενθουσιώδη περίοδο οποίων μας υπό τη δική σας ε, προεδρία, πρόεδρε, και η κυρία Κεσλέρα αναφέρθηκε στο θέμα του Ευρωπαϊκού Μεσολαβητή. Εγώ πάντοτε είμαι μυστικοπαθής, αλλά τώρα θα σας αποκαλύψω ένα μυστικό ότι εγώ είμαι κατά της ιδέας του διαμεσολαβητή, γιατί πιστεύω σε λιγότερη δημοκρατία και όχι σε περισσότερη. Γιατί επανεφευρίσκουμε κάτι όταν έχουμε ήδη το μηχανισμό και σίγουρα δεν θέλω ένα διαμεσολαβητή, ο οποίο θα μπορούσε εν δυνάμει να έρθει σε σύγκρουση με την ε, λήψη αποφάσεων. Να έχουμε λοιπόν λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη βοήθεια προ την ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να φτάνει και που πρέπει. Ευχαριστώ. Κύριο Μέσνερ. Ich würde gerne noch mal die Frage des για το θέμα της ε, γενικότερης έτσι, ιστορίας, να πω κάτι. Ο Επίτροπος ανέφερε ότι η μεγαλύτερη, διακυβέρνηση, η μεγαλύτερη ε, πρόκληση είναι η διακυβέρνηση. Όλοι από, την, ε, από το Think Tank συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Αλλά αυτό που θέλουμε να προσθέσουμε στο, στη δική μας προσφορά είναι ότι αυτή η διακυβέρνηση θα πρέπει να συνδυαστεί με την συμβολή της αναπτυξιακής πολιτικής, των παγκόσμιων προκλήσεων και της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Μετανάστευση, διασυνοριακές συγκρούσεις, κλιματικές αλλαγές, δημογραφικές αλλαγές, απώλεια πόρων, αντιμετώπιση της φτώχειας, αξιο, αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Είναι θέματα γενικά. Και επίσης πρέπει να δούμε το πράγμα και από την πλευρά των προκλήσεων που δεν μπορούν όμως να λυθούν χωρίς την ε, βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι προς κοινό συμφέρον όλων μας λοιπόν να λυθούν. Τώρα, πώς θα θέσουμε προτεραιότητες. Το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Ο Επίτροπος πολύ σωστά λέει ότι αν διαβάσει κανείς τον, ε, το ε, βιβλιαράκι αυτό, έχει έναν μεγάλο κατάλογο με πολλές προτεραιότητες και πολλές προκλήσεις. Τι γίνεται λοιπόν. Φοβούμε ότι η απάντησή μας είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να, να ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα αυτά από ευρωπαϊκή πλευρά, εάν θέλουμε να μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο. Ίσως αυτή είναι η απάντηση, γιατί η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι να θα πάρουμε μία από αυτές τις 3, 4, 5, 6 προκλήσεις, μετανάστευση ας πούμε, ή ε, έλλειψη, έλλειψη πόρη, ως Ευρωπαϊκή, ως, Ευρωπα... ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί στη συμβολή μας. Αρκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Καμία... Κανένα από τα, κράτη, από τα μελη μας δεν μπορεί να το λύσει μόνο το, το πρόβλημα αυτό. Ούτε ένα. Γι' αυτό είναι σημαντική η Ευρώπη και γι' αυτό το θέμα είναι πώς μπορούμε να επιτύχουμε να, συνδε... να συνδυάσουμε όλες τις προσπάθειες. Και νομίζω ότι αυτή είναι η απάντησή μας. Δεν θα καταλήξουμε στο να λέμε ότι ω Ευρώπη θα επικεντρωθούμε σε ένα ή σε δύο, σε μία ή σε δύο προκλήσεις. Όχι. Η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί με όλα τα θέματα αυτά και να συμβάλλει αποτελεσματικά σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω προς τους εμπειρογνώμονες μας. Έχετε μετρήσει τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που έχουν χαθεί στην Αφρική λόγω της αλληλευτικής μας πολιτικής. Μπορεί εδώ η εμπειρογνώμονας ε, της ε, αλληλευτική πολιτική θα μπορούσε να σα το πει. Γνωρίζετε λοιπόν τον αριθμό αυτών των θέσεων απασχόληση που χάθηκαν. No. I think that Isabel should then... Η Ισαμπέλ μπορεί να σας διαφωτίσει. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία, αλλά είναι γεγονός ότι έχει συμφωνίες ε, εταιρική σχέσης αλλιευτικές με μερικές χώρες της Δυτικής Αφρικής, ε, με αρκετές χώρες της Δυτικής Αφρικής. Οι συμφωνίες αυτές ε, από το 2002 προβλέπουν ότι ένα τμήμα ε, των χρημάτων ε, που ε, λαμβάνονται για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλιεύει στα ύδατά τους πρέπει να πηγαίνει στην υποστήριξη της τοπικής, του τοπικού αλλιευτικού κλάδου. στη Σενεγάλη, στη Μαυριτανία, στη Γουινέα Μπισάου. Ε, μπορεί λοιπόν να υποστηριχθεί η τοπική κοινότητα των αλλιέων μόνο αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλιεύει. Και ποια είναι η ηρωνία. Ότι Ουσιαστικά υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ της τοπικής κοινότητας και των ε, ευρωπαϊκών ε, σκαφών και δεν, υπάρχει καθόλου, δεν υπάρχουν στατιστικές σε αυτές τις χώρες, ε, κυρία Πρόεδρε, των ανθρώπων που έχουν την αλληλεία ως βασική πηγή εισοδήματος. Ε. Στη Σενεγάλη, για παράδειγμα, 600.000 άνθρωποι έχουν την αλεία ως βασική πηγή εισοδήματος και τα αποθέματα έχουν μειωθεί εν μέρη εξαιτίας αλληλευτικής δραστηριότητας των, σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ως φορολογούμενοι ουσιαστικά επιδοτούμε πλειοκτήτες αλλιευτικών σκαφών για να αλλιεύουν σε αυτές τις χώρες. Γιατί η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει μια εξωτερική διάσταση και η εξωτερική διάσταση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τρόφιμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα, 20% του προπολογισμού της κοινή αλληλευτικής πολιτικής πηγαίνει στις εξωτερικές, ε, σε αυτές τις συμφωνίες εξωτερικές, ε, τις εξωτερικές ε, και δεν ξέρω τελικά Η πραγματική αναπτυξιακή πτυχή θα ήταν να βοηθήσουμε την ύπαρξη υποδομής στις χώρες αυτές, ώστε να μπορούν να εξάγουν ψάρια στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα στις ε, πολιτικές που θα έπρεπε να βάλει τάξη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να μην είναι πολύ κοινική η προσέγγιση μου. Πώς λοιπόν, λέει η Πρόεδρος, μπορείτε να μιλάτε για δημιουργία θέσεων απασχόληση, αν δεν έχετε λάβει υπόψη τις εκατοντάδες χιλιάδες καμένων θέσεων εργασίας λογικό, Κοιτάξτε, δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα όταν μιλάμε για ανάπτυξη. I'm the president of this. I shouldn't take the floor myself. So. I think that... Λοιπόν, είμαι η πρόεδρος, ε, αλλά και εγώ μερικές φορές θέλω να παίρνω το λόγο, ο κύριος Γκέρενς. Έχω τρία-τέσσερα σχόλια για το συντονισμό καταρχήν. Ε, δεν ξέρω αν το συζητήσατε προηγουμένως, αλλά έχουμε το 80% της βοήθειας που δαπανάτε από τα κράτη-μέλη. Ενώ η συνθήκη της Λισαβόνας ε, προβλέπει την εισαγωγή της αρχής του συντονισμού των αναπτυξιακών ε, πολιτικών έτσι λοιπόν έχουμε τα 27 κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 28 πρωταγωνιστές, ενώ εδώ ε, είναι σαν να μιλάμε για όλη την αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ το ουσιαστικό κομμάτι της αναπτυξιακής βοήθειας το διοχετεύουν τα κράτη-μέλη. Ποιος το σκέφτεται αυτό και ποιος κάνει αυτό το συντονιστικό έργο. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Τώρα δεύτερη παρατήρηση για το συντονισμό. Αναφερθήκατε στην πρόθεση της διακυβέρνησης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολύ ωραία, πρέπει να γίνει αυτό. Όμως, ε, δεύτερον, θα πρέπει να σκεφτούμε και κάποια διάρθρωση ε, στην απάντηση που θα δοθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις. Βλέπουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει μια καθολική επισκόπηση των πραγμάτων στο νομισματικό τομέα, όπου ε, στον εμπορικό τομέα η ΔΟΕ που κάνει ακαδημικό έργο περισσότερο γιατί περισσότερο το έργο αυτό υλοποιείται στις διεθνείς συνεδριάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο να ρυθμίζει τις διαφορές που μπορεί να προκύπτουν. Τι προτείνεται λοιπόν ως ε, γέφυρα μεταξύ αυτών ε, των θεσμών, μεταξύ αυτών των οργάνων και τι πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχει μεγαλύτερο βάρος με μία μόνη φωνή στο διευθυντικό Ταμείο, στον ΠΟΕ και σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα. Και τρίτο σχόλιο, αρχίζει να με ενοχλεί κάτι. Δεν ακούω σχεδόν καθόλου τη λέξη εταιρική σχέση ούτε ενδογενή ανάπτυξη. Οι συνομιλητέ μα στην Αφρική, όταν μιλάμε για τη Γεωργία, είναι η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συνδικάτων. Ε, όταν ε, ε, μιλώ με τους αρμόδιους για την αγροτική πολιτική, ακούω μία συγκεκριμένη διάρθρωση λόγου, ενώ όταν μιλάμε με τους υπουργούς οικονομικούς ακούω ένα διαφορετικό λόγο. Τελικά, ποια είναι η βούληση των λαών και τι επιλέγουμε εμείς, τι συγκρατούμε ως βούληση των λαών. Η ενδογενής ανάπτυξη είναι ε, ουσιαστικά κάτι πολύ σημαντικό. Ένας ε, μεγάλος Αφρικανός σοφός, ο είπε ότι στην, ε, στην Αφρική αναπτυσσόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στην ενδογενή ανάπτυξη, γιατί εγώ νομίζω ότι αν μιλάμε για ανάπτυξη μόνο, έχουμε μία βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Αν έχουμε μικρόπιστοση, ε, τελικά βλέπετε ότι ε, έχουμε επιστροφή 300% του αρχικού κεφαλαίου ενώ αν δανείσει κανείς επίπεδο κράτους, από κράτος σε κράτος ε, δεν επιστρέφεται ούτε ένα ευρώ. Τελικά μιλάμε για κύρωση του χρέους, για διαγραφή του χρέους ε, και ποτέ δεν έχουν επιστραφεί κονδύλια και αυτά που δεν έχουν επιστραφεί ποτέ μάλλον θα χρησιμοποιηθούν για να παρουσιαστούν ως δημόσια για βοήθεια στην ανάπτυξη. Ε, Ούτω ή άλλω αυτά τα χρήματα ποτέ δεν επιστρέφουν στο Ταμείο του Κράτου ε, και φυσικά αυτό φουσκώνει τον αριθμό τη ε, βοήθεια για την ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο θέμα τη αποτελεσματικότητα. Δεν διάβασα όλο το εγγραφό σα, ε, τώρα το ανακάλυψα, αλλά θα ήθελα να μπορέσετε να λάβετε υπόψη αυτέ τι παρατηρήσει. Λοιπόν, έχω και μια ακόμα ερώτηση για τους εμπειρογνώμονες. Γνωρίζετε τη σχέση μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και των παράνομων ροών που βγαίνουν, έκρογων μάλλον, από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γνωρίζετε τη σχέση αυτή. Πόσα ήταν. Uh, so, uh, σαν φορέ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε όταν μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια. Πραγματικά εδώ βλέπουμε ότι το σύστημα από την αρχή από την χάνει να λειτουργήσει. Η κυρία Τσίμερ έχει ζητήσει το λόγο. Σύντομα. Ήδη πολλά ερωτήματα ετέθησαν ήδη, τα οποία σχετίζονται πολύ πιο συγκεκριμένα στην, ε, με, την, ε, με το βιβλιαράκι αυτό. Θα ήθελα να σας ευστήσω την προσοχή σε κάτι. Προσπάθησα το χρόνο που έμεινε να δω ποιες είναι οι συστάσεις σας, έτσι, να καταλάβω γενικά. Και συμφωνώ γενικώ με τους προσδιορισμούς που, έχετε θέσει και όντως ε, πρέπει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων πολιτικής και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να εφαρμοστούν ε, ώστε να έχουμε και μια αποτελεσματική πολιτική γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε την ε, κρίση που περνάει ο πλανήτης. Αλλά τον τελευταίο καιρό, ακριβώς στο σημείο αυτό, η παγκόσμια κοινότητα αρνείται να δράσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανταποκριθεί στο ρόλο της ως, ε, ως ε, ε, παγκόσμιο παίχτη. Ε, στην Κοπεχάγη, ας πούμε. Ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Ειδικά σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, τον αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τη σύνδεση με την αντιμετώπιση της φτώχεια και την εφαρμογή των ε, στόχων της χιλιετία. δεν, αρθ, δεν ε, ε ήρθε στο, στο ύψος των ασέων. Οπότε, με την ε, ε στρατηγική για το 2020, αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί σε ό,τι αφορά ότι είναι παγκόσμιος παίχτης. Νομίζω ότι πρέπει πολύ συγκεκριμένα να θέσουμε το θέμα αυτό και θα πρέπει, πρέπει πραγματικά να επηρεάσουμε τα πράγματα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Γιατί αυτό εδώ που προτείνετε εσείς και αυτό που ζητάτε ε, γίνεται, καθίσταται αδύνατο. Είναι αδύνατο να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Τουλάχιστον η δική μου εντύπωση είναι αυτή μέσω των προσεγγίσεων που προτείνεται. Δεν αντικατοπτρίζονται τα πάντα εδώ. Πώς λοιπόν θα καταφέρουμε να αποτελέσει αυτό τη βάση των πολιτικών και στρατηγικών εξελίξεων και καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα που προκύπτει από αυτό το κείμενο που διάβασα. Ευχαριστώ. The 10 λεπτά μας δίνουν οι διερμηνείς, το πολύ. We should share this time between ο κύριος Έγγελ και ο κύριος Γιούγκ θα μοιραστούν αυτά τα δέκα λεπτά για να απαντήσουν. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ανησυχίες που ακούσατε. Κοιτάξτε, πολύ θα το ήθελα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου ετέθησαν. Το ζήτημα της διακυβέρνησης ετέθη σαφώς νομίζω και θα ήθελα μία παρατήρηση να κάνω ότι στη μας, ε, κατά τη δική μας άποψη και μιλάω για το δικό μας ε, πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EuroPaid έχουν εξελιχθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ε, μιας προσέγγισης διακυβέρνησης εντός της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζεται. Και αυτό τι τεράστια πρόκληση της κατανομής εργασιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι να λέμε αφήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό στο οποίο είναι καλύτεροι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ε, γίνεται η κατανομή. Και απαντώ σε αυτό που είπε για τις ε, διμερείς συμφωνίες η κυρία Κέλλερ. Καλή είναι οι διμερείς δωρητές μερικέ περιπτώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλή σε άλλα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτό το ποιοτικό άλμα ως προς την ε, βοήθεια ε, της αναπτυξιακής, ε, την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τη δημιουργία πλούτου, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρον το παράδειγμα για την αλληλεία. Είναι ελάχιστο εμπόδιο στα προβλήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν μιλάμε ακόμη για την κοινή αγροτική πολιτική, δεν μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, δεν μιλάμε για την ε, διαδικασία ε, ΙΠΑ. Γι' αυτό νομίζω ότι ζητήματα υπάρχουν πολλά και γι' αυτό ακριβώς δίνουμε τόση ιδιαίτερη, τόση σημασία ε, στην ε, πολιτική της αναπτυξιακής βοήθειας ε, και τη συνοχή της. Δεν είναι όπως μας ρωτάνε για παράδειγμα τι, κάνετε, τι κάνετε για την ανάπτυξη και λέμε α, ό,τι κάνουμε είναι συμβατό με την εξωτερική πολιτική. Μιλάω για τη συνοχή της πολιτικής ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και σημαντικός παράγοντας αν θέλει κανείς να έχει καλή κατανομή εργασιών και μια ενιαία φωνή για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της ανάπτυξης και όχι κατά αυτής. Επίσης, το ερώτημα, πολύ θεμητό, είναι τι μπορούμε να κάνουμε στις χώρες εταίρους, στις αντιπροσωπείες, ώστε να υπάρχει περισσότερη παρακολούθηση ε, για την έλλειψη συνοχής να εντοπίζεται δηλαδή το πρόβλημα. Γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με την ε, συνοχή της πολιτικής είναι ότι έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση γιατί υπάρχουν τόσες πολλές, ε, υπάρχει πολλή έρευνα, μιλάμε για την κοινή γεωργική πολιτική, την γνωρίζουμε και την κοινή αλληλευτική πολιτική. Αλλά έχουμε κάνει μόλις ε, τις τρεις πρώτες μελέτες για, για συγκεκριμένες χώρες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν υπάρχει κόσμος επιτόπου να εντοπίζει ακριβώς ε, τις ε, ασυνέπειες, δεν γίνεται τίποτα. Για να υπάρξει λοιπόν αυτή η δυνατότητα του feedback για τις ε, ασυνέπειες, δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στις ιδιωτικές εταιρείες και στις μικρομεσαίες, συγγνωμικές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για το συντονισμό. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν μπορεί επιτυχώς να συντονίσει τον εαυτό της, το είπε νομίζω και ο Επίτροπος, ε πώς θα πάμε να διακηρύττουμε εμείς συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει επιτέλους να πούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορούμε να έχουμε χιλιάδες δωρητές ε, εκ μέρου μα. Πρέπει κάπως να τα περιορίσουμε τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε πιο εστιασμένοι, καλύτερη κατανομή εργασιών. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό με πολιτικό τρόπο. Και αυτό νομίζω, νομίζω ότι εδώ είναι το φόρουμ που μπορεί να συμβεί αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, εγώ για να πω για την ατζέντα τη διακυβέρνηση, δεν είναι θέμα να δαπανίσουμε τεράστια επιπρόσθετα ποσά. Συνήθω δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα μέσω τη πρωτοβουλία για τη διακυβέρνηση, μέσω διμερών πρωτοβουλειών, Δεν έχουμε πολύ χρήματα εκεί όπου δεν βελτιώνονται ή επιδεινώνονται οι δείκτε για τη διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε το θέμα ε, της ε, πολιτικής μεταρρύθμισης μαζί με το τοπικό ownership. Θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει από έτοιμα από τα μέσα και θα έλεγα ότι πρέπει πραγματικά να δούμε ποιος είναι ο πολιτικός αντίκτυπος της δημοσιονομικής στήριξης. Ξέρουμε ότι οι δωρητές ε, ουσιαστικά προβαίνουν σε χρηματοδότηση μέσω της ε, άμεσης ε, στήριξης, όμως δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος στην τοπική πολιτική δυναμική. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί, το χάρη, να έχουμε επιδίνωση της διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας. Τέλος, η Κομισιόν μας ε, ρώτησε μήπως ε, βάζουμε πάρα πολλά στοιχεία στην εξίσωση. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα εκτροπής ε, πόρων από κύριους, από κύριες προκλήσεις ανάπτυξη όπως είναι τα κράτη η ασφάλεια και η ειρήνη, αλλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλα τα μέσα μας έτσι ώστε να ε, χορηγούμε πιο αποτελεσματικά τη βοήθεια. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό πίεσης ομοτήμων όπου μπορούμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα μέσα που έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στη δυναμική σειράξεων, στη δημιουργία πλούτου έτσι ώστε να ασκήσουμε κάποια μόχλευση επί πολιτικών που έχουν επιζήμιο αντίκτυπο βλέπετε εδώ ότι πρέπει να ε, υπάρχει και συνέπεια με την πολιτική εμπορίου. Το παράδειγμα με το Μαρόκο είναι, ε, ε μας δείχνει πάρα πολλά ε, ο ευρωπαϊκός προστατευτισμός στον τομέα της γεωργίας για το Μαρόκο ε, έχει 5 ή 6 φορές, είναι 5 ή 6 φορές μεγαλύτερη η 6 φορες ειναι πέντε η 6 φορες μεγαλυτερη η ζημια σε σχέση με τη βοήθεια που δίνουμε. Τώρα αν μιλήσουμε για την ε, πρόσβαση στο GSP. Πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο έχει στον κατακαιρματισμό της χώρας. Το G20 ήδη, έγινε, ε, ήδη δόθηκε μία υπόσχεση στο ότι πρέπει να ε, δώσουμε μία έμφαση στη σκοπιά της ανάπτυξης καταπολεμώντας τον προστατευτισμό. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό που θα μπορούσε να αποκαλύψει αυτές τις συνέπειες και να ασκηθεί πίεση στα κρατημέλη. Αυτό ήταν πολύ ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα προς τα μπρος. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συνεισφορές σας. Όλα αυτά ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα για μας. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Έτσι λοιπόν, ε, να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, ε, στις 22 Μαρτίου από τις 3 ε, ως τις 6.30 ε, και στις 22 ε, Απριλίου από τις 3 ως τις 6.30. Εδώ ολοκληρώνουμε τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους να καταλήψετε αμέσω στην αίθουσα και να συνεχίσετε τη συζήτησή σας εκτός της αίθουσας αυτή, γιατί χρειαζόμαστε την αίθουσα αυτή για μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών μεταξύ των συντονιστών μας και του Επιτρόπου Πίμπλεξ που θα ξεκινήσει τώρα. Οι μόνοι που θα παραμείνουν στην αίθουσα τώρα είναι ο Πίτροπος Πίμπαλξ, τα μέλη του γραφείου του, ε, τα πέντε μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής μας και οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων, αλλά όχι ε, οι αναπληρωτές ε, ή η βοηθή ένας μόνο υπαλλήλο από κάθε πολιτική ομάδα και τρία άτομα από τη γραμματεία, ο βοηθός της Κομισιόν, Καλό λοιπόν όλου του υπόλοιπου να εγκαταλείψουν την αίθουσα αμέσως και καλό το κλητήρα να ε, διασφαλίσει ότι κανείς από όσου δεν αρμόζουν θα παραμείνει στην αίθουσα για την ε, επόμενη συνάντηση.